Κυρίε και κύριοι, καλημέρα σας. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε, ε, διότι ήδη έχει περάσει λίγο η ώρα. Έχουμε σήμερα ένα πολύ σημαντικό θέμα προς συζήτηση και έχουμε έγγραφα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία ανέλαβε να μας παρουσιάσει ε, το θέμα των ε, πυρηνικών αποβλήτων και την διαχείρισή τους ως συνήθως και αυτό δεν είναι καινούριο έχουμε ένα πολύ πιεσμένο πρόγραμμα αλλά θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε σωστά το χρόνο μας γι' αυτό και χωρίς πολλά πολλά δίνω το λόγο εις τους συναδέλφους με τους οποίους πρόκειται να έχουμε τις τεχνικές συζητήσεις όπως άλλωστε το λέει το πρόγραμμα καταρχήν θα δώσω τον λόγο στον κύριο Ριώτε ο οποίος είναι επικεφαλής ε, στον ε, ΩΣΑ για την ε, προστασία από ακτινοβολίες και τη διαχείριση των πυρνικών αποβλήτων και του δίνω το λόγο κατευθείαν. Καλημέρα σας κύριε και κύριοι, χωρίς μικρόφωνο όμως. Μικρόφωνο. Παρακαλώ. Τώρα μάλιστα. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω διάφορες απόψεις και αποτελέσματα του, ε, ε, ε, του γραφείου του ΟΣΑ για την πυρηνική ενέργεια και στο θέμα αυτό θα ήθελα να κάνω μία σύντομη παρουσίαση του ΩΣΑ για να ξέρετε περί τίνος ομιλούμε και μετά θα πω μερικά πράγματα ε, για την ε, ε, διαχείριση των αποβλήτων και θα αναφερθώ και σε διάφορα θέματα τα οποία νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να συζητάμε σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Ε, ο ΩΣΑ έχει 33 μέλη, είναι η τελευταία, ε, ο τελευταίος απολογισμός και ίσως και η Εστονία προσχωρήσει σε λίγο και μέσα στο 2012 η Ρωσία βέβαια ε, δεν συμμετέχουν οι ασυνοί, ε, δηλαδή όχι όλες οι πολιτικές ομάδες, αλλά ελπίζουμε ότι μέχρι τον Απρίλιο του χρόνου θα υπάρξουν αλλαγές. Βεβαίως ε, είμαστε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με την IEA στη Βιέννη και η ουσιαστική εργασία δεν γίνεται από τη γραμματεία αλλά από τις ομάδες εμπειρογνώμων Έχουμε ε, πολλούς ε, εμπειρογνώμονες. Κάτι συνέβη αλλά θα προσπαθήσω να συνεχίσω. Έχουμε 1.500 ειδικού και η εργασία μας είναι ουσιαστικά εργασία των εμπειρογνωμόνων διεθνώς. Και με αυτό Εννοώ ότι τα αποτελέσματα της εργασίας μας έχουν, είναι υψηλού επίπεδου και έχουν κύρος. Ε, αποβλέπουμε δε στην αμοιβαία κατανόηση. Επίσης πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ένα μείγμα των διαφόρων ειδικοτήτων και το θέμα της διαχειρίσεως των αποβλήτων συνεργαζόμαστε με, ήδη με τη Ρουμανία, την ε, Σλοβενία και τη Ρωσία ε, και βεβαίως ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση όπου έχουμε και έναν εκπρόσωπο ε, όσον αφορά την, ε, ε, τον οργανισμό πυρηνικής ενεργείας πρέπει να τονίσω ότι υπάρχει και ένα γραφείο το οποίο ασχολείται από 10 χρόνια με τις επιπτώσεις για την κοινωνία. Οπότε τώρα θα ήθελα να αναφερθώ στην ισχύουσα κατάσταση διότι θεωρούμε ότι ε, υπάρχει, ε, υπάρχουν διάφορα ε, σημεία όπου μπορεί κανείς να αποθέσει τα πυρνικά απόβλητα και υπάρχει ένας κύκλος για αυτά τα σημεία εναπόθεσης χωρίς βέβαια να συμπεριλαμβάνουμε τους τύπους των για όλους τους τύπους των πυρηνικών αποβλήτων που δεν προκαλούν θερμότητα. Υπάρχουν δε ορισμένες χώρες οι οποίες θέλουν να έχουν σημεία εναπόθεσης ε, βαθιά στο έδαφος και ε, το πιο χρήσιμο είναι να κοιτάξουμε συγκεκριμένα θέματα όπως ε, τα μικρά, μικτά απόβλητα, γραφίτες κτλ. Ε, υπάρχουν ε, και διάφορα απόβλητα τα οποία θεωρούνται ε, εξωτικά και, δύο και δυνατότητα για εναπόθεση σε εξωτικά σημεία ε, ε, υπάρχουν όμως ε, θέματα ασφαλείας που πρέπει να ληφθούν υπόψη και βεβαίως η μεταστοιχείωση είναι κάτι που μας απασχολεί και σαν ε, μακροπρόθεσμη λύση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε τώρα και θα επανέλθω στο σημείο αυτό. Άλλωστε ε, και ο κύριος Στομάσκι θα συζητήσει το θέμα αυτό για τους προχωρισμένους ε, κύκλους καυσίμων και την μεταστοιχίωση, διότι ε, θεωρούσαμε ότι άμεσα έχουμε μία μείωση του όγκου αλλά υπάρχουν και πρέπει να υπάρχει ε, σημαντική επίπτωση για τον όγκο για την θερμότητα των αποβλήτων και ε, αυτά μπορούν να επιτευχθούν μόνο σε πλήρως κλειστούς κύκλους καυσίμων χρησιμοποιώντας αντιδραστήρες υψηλής ταχύτητος. Άρα αυτό είναι κάτι που πρέπει να σκεφτούμε για το μέλλον αλλά δεν είναι κάτι που θα λυθεί από τη μια μέρα στην άλλη. Επίσης όσον αφορά την εναπόθεση, ε, πολλές ε, φορές ε, η permanent stewardship δεν είναι δυνατή και σε αυτή την κοινότητα υπάρχει μία συμφωνία, πρέπει δε να υπάρχει επιστημονικά και τεχνικά μία μακροπρόθεσμη λύση. Γι' αυτό και έχουμε δημοσιεύσει συλλογικές γνωμοδοτήσεις ε, για το πώς θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στην διάθεση των γεωλογικών αποβλήτων με πλήρη προστασία και με τεχνικά εφικτές δυνατότητες. Πρέπει όμως από την αρχή να συμμετάσχουν και οι ενδιαφερόμενοι και θα δείτε ότι υπάρχουν διάφορες εναλλακτικές λύσεις σε διάφορα κράτη αναλόγως του πολιτικού πλαισίου της ε, κάθε χώρας και περιοχής αλλά υπάρχουν ουσιαστικά κοινοί στόχοι όσον αφορά την ασφάλεια και το ζητούμενο στόχο. Οπότε τώρα έχουμε πολύ περισσότερες πληροφορίες και τουλάχιστον ένα πρόγραμμα μπορεί να καταρτιστεί για όλες τις χώρες που έχουν τέτοιου είδους απόβλητα. Πολύ σύντομα θα ήθελα να αναφερθώ σε ποιους τομείς ε, εξετάζουμε και αντιμετωπίζουμε από κοινού και να δούμε και ποιες είναι οι μακροπρόθεσμες σχέσεις. Υπάρχουν ε, συνθήκες ε, που διέπουν τα θέματα αυτά. Έχουμε και συστάσεις της ICRP. Ε, εάν λοιπόν ε, ε, δούμε τις συστάσεις αυτές θα δούμε ότι υπάρχουν ουσιαστικά κοινοί κανόνες στις περισσότερες περιοχές αλλά οι μέθοδοι είναι διαφορετικοί που χρησιμοποιούνται στις διάφορες χώρες και δεν υπάρχει και ο, ίδιος βαθμός οριμότητος. Γι' αυτό και πρέπει να δούμε πώς μπορεί να ρυθμιστεί η μακροπρόθεσμη ασφάλεια διότι ορισμένα κριτήρια χωρών αναφέρονται στους αριθμούς του κινδύνου σε άλλους όλους στο χρονικό πλαίσιο και στις ε, ε, αξίες. Ε, είδαμε ότι τα θέματα αυτά έχουν εξεταστεί από την αρμόδια επιτροπή και μπορέσαμε να διαπιστώσουμε ότι έτσι μπορεί να καταλήξει κανείς σε ένα ε, υψηλό επίπεδο ασφαλείας για τους ανθρώπους αλλά υπάρχουν και ορισμένοι παράγοντες ε, αμφιβολίας όσον αφορά τα κριτήρια αυτά. Ε, τεχνικά θέματα, τεχνική εμπιστοσύνη η οποία δεν θεωρείται γενικώ σαν ένα ε, σοβαρό πρόβλημα διότι πιστεύουμε ότι μπορεί να ισχύσει για όλους, για τα προγράμματα τα οποία ε, χρησιμοποιούνται και εμφανίζουν το πώς ε, έχει η κατάσταση ε, και από πλευράς ε, ασφαλείας είναι πολύ σημαντικό να μην αναφερόμαστε μόνο στα αριθμητικά αποτελέσματα των προγραμμάτων υπολογιστών αλλά να έχουμε και δείκτες οι οποίοι δεν είναι εύκολο να μεταφραστούν με ακρίβεια σε αριθμούς. Αυτό που είναι επίσης σημαντικό είναι το, η εργασία που γίνεται εις ε, ε, τα εργαστήρια και δεν πρέπει να υποβαθμίζουμε τον ε, ρόλο των αρχών εποκτείας που ισχύουν σε όλες τις χώρες που έχουν κάποιο πρόγραμμα και επίσης και τις ε, μελέτες που καταρτίζουν οι ομολογοί μας. Ε, υπάρχει μεγάλη, ε, μεγάλο ενδιαφέρον για περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη και σχετικά προγράμματα για τις σύγχρονες μεθόδους κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την έρευνα και ανάπτυξη ακόμη και όταν ήδη εφαρμόζουμε και δημιουργούμε τα σημεία εναπόθεσης. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να αναφερθώ σε ορισμένες δραστηριότητες. Έχουμε ένα φόρουμ εμπιστοσύνης των ενδιαφερομένων ε, για περιοχές ε, οι οποίες λαμβάνονται ε, υπόψη σαν σημεία εναποθέσεως στη Φιλανδία, στον Καναδά, στο Βέλγιο, στη Γερμανία, στην Ισπανία, στην Ουγγαρία, στη Γαλλία και στη Σουηδία για το 2011. Υπάρχει γενική Ευρωπαϊκή Αρχή ε, για ε, συμμετοχή των ε, ενδιαφερομένων οι οποίοι όμως θα πρέπει να έχουν κοινέ αξίες και στόχους σχετικά με το θέμα αυτό. Χρειαζόμαστε λοιπόν πέραν των τεχνικών αδειών και μία κοινωνική νομιμοποίηση του συστήματος αυτού και γι' αυτό πιστεύω πιστεύουμε ότι τα προγράμματα θα πρέπει ε, να προχωρούν ε, βαθμιαία και να μπορούν ε, να ε, προχωρήσουμε ή να αλλάξουμε πορεία αναλόγως ε, της αξιολογήσεως ή σε ορισμένα σημεία να οπισθοχωρήσουμε. Οπότε για να ισχύσει αυτή η διαδικασία πρέπει να υπάρχουν διάφανες διαδικασίες και δυνατότητα συμμετοχής όλων και θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι από πλευράς του κοινού η διαδικασία είναι πολύ σημαντική και ε, είναι εξίσου σημαντική όσο και το αποτέλεσμα αυτής της ε, διαδικασίας αξιολογήσεως. Ένα βασικό θέμα προσυζήτηση τώρα και που ε, θα προκύψει και στο μέλλον είναι η της και η και ο τρόπος επανακτήσεως μιας ε, ε, ε, ενός προϊόντος από το σημείο εναποθέσεως διότι αυτή τη στιγμή ε, δεν ε, ε, έχουν όλοι συμφωνήσει για την σκοπιμότητα των υπογείων σημείων εναπόθεσης άρα υπάρχει αλλαγή της αντιλήψεως σχετικά με αυτά τα σημεία εναποθέσεως. Βεβαίως όλα αυτά είναι ε, πάντοτε ε, εξετάσιμα και υπάρχουν και ε, διακοιμάνσεις δηλαδή δεν μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα θέματα με μία κοινή λύση για όλοι λύση η οποία θα μπορούσε να στηριχθεί ε, διότι θα έπρεπε να προχωρήσουμε και να μην περιμένουμε να δούμε τι μελγενέστε στο τέλος και τέλος θα ήθελα να αναφερθώ σε μία μελέτη την οποία κάναμε πρόσφατα που είναι πολύ σημαντική και έχουμε διατυπώσει πρότυπα συνεργασίας για την περιοχή ε, και ε, για τις ε, τα γραφεία τα οποία εφαρμόζουν αυτά τα μέσα ε, διότι ο τρόπος με τον οποίο προχωράμε είναι ότι δίδουμε κάποια δικαιώματα εις ε, την ε, κοινότητα και βεβαίως στη συνέχεια θα έπρεπε να υπάρχει και το δικαίωμα αποσύρσεως σε κάποιο σημείο. Είναι σαφές ότι αυτή η συνεργασία πρέπει να στηρίζεται με ορισμένα μέτρα και ιδίως οι κοινότητες να δεχθούν να στεγάσουν αυτά τα σημεία εναπόθεσης και ε, αυτό μπορεί να γίνει ε, είτε με μεγαλύτερη στήριξη εκ των έξω είτε με εκπαίδευση των ενδιαφερομένων υπάρχουν δε ε, και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα προσόντα ιδίως όσον αφορά την ποιότητα ζωής των ενδιαφερομένων θα ήθελα να σας αναφέρω εδώ ένα συνέδριο το οποίο θα γίνει στην Ιαπωνία του χρόνου τον Οκτώβριο που αναφέρεται τα γεωλογικά σημεία εναπόθεσης. Είναι ε, ένα συνέδριο που διοργανώνεται ανά τετραετία και ε, αναφέρουμε ποια είναι τα θέματα για τα ε, σημεία αυτά εναπόθεσης και όπως σας είπα είναι θέματα εμπιστοσύνης και περιφερειακής στηρίξεως. Θεωρούμε ότι τεχνικά αυτή η λύση είναι εφικτή και μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορες συνθήκες. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα τα οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη. Ε, αισθανόμαστε ότι υπάρχει ε, τεχνική εμπιστοσύνη η οποία βασίζεται ή στην ε, συνεργασία. Υπάρχει μία λήψη αποφάσεως, μία διαδικασία λήψης αποφάσεων η οποία στηρίζει την προσπάθεια και γνωρίζουμε ότι υπάρχει ε, πάρα πολύ μεγάλη πείρα για να οργανωθούν προγράμματα ε, για τους ε, εντόπιους ενδιαφερόμενους και γι' αυτό οργανώνουμε διάφορα συνέδρια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ε, θαυμάσια παρουσίαση και τις πληροφορίες που μας δώσατε και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Τομάουσκε ο οποίος είναι ε, επικεφαλής ε, του τμήματος κύκλου πυρνικών καυσίμων στο Πανεπιστήμιο του Άχεν. Ευχαριστώ κύριε Ρόιλ. Θα ξεκινήσω πάρα αυτά. Μόλις ε, ετοιμαστούν οι διαφάνειες, θα μιλήσω για την μεταστοιχείωση ως εναλλακτική λύση για τη διαχείριση των ε, πολύ ραδιενεργών πυρηνικών αποβλήτων. Καταρχάς, θέλω να πω δύο λόγια για την πυρηνική έρευνα και την ε, εκπαίδευση που κάνουμε στο Άχεν για τη μεταστοιχείωση ε, ο λόγος είναι η μείωση της ραδιενέργειας των ε, πολύ ραδιενεργών ε, αποβλήτων. υπάρχει το πολιτικό πλαίσιο στη Γερμανία, η τελική διάθεση, η έννοια, η σύλληψη του αγκάτε. Δύο λόγια για τη μελέτη σκοπιμότητας, για την έννοια της μεταστοιχίωσης που έχουμε κάνει ή κάνουμε, εξακολουθούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή και θα κάνουμε μια σύγκριση μετά με την ε, βελγική ε, μεταστοιχείωση, το πρόγραμμα ΜΥΡΑ, τα επόμενα στάδια, μετά θα για τα επόμενα στάδια και μετά ε, τα συμπεράσματα. Καταρχάς, η εκπαίδευση και η έρευνα. εγώ ανήκω στο Ινστιτούτο, Κύκλου των Πυρηνικών Καυσίμων στο Άχεν και υπάρχει αυτό το Ινστιτούτο από το 2008 στο Πανεπιστήμιο του Άχεν. Ε, αναπτύσσουμε ε, καινοτόμες τεχνικές λύσεις για όλο τον κύκλο ζωής του πυρηνικού καυσίμου και μετά από 1,5 χρόνο έχουμε 25 υπαλλήλους σε 4 ομάδες εργασίας. Επίσης υπάρχει ένα άλλο Ινστιτούτο στο Άχεν ε, για την ασφάλεια του αντιδραστήρα και για την τεχνολογία του αντιδραστήρα υπό την αιγίδα του συναδέλφου του κ. Αλελάιν. Ε, η έρευνα καταρχάς. Έχουμε καταρχάς το θέμα της ε, πυρηνικής ε, προμήθειας και της διάθεσης. Κάνω μια ανάλυση της ασφάλειας των προγραμμάτων ε, εναπόθεση στη Γερμανία, εν συνεχεία μεταστοιχείωση και χαρακτηρισμός των ραδιενεργών αποβλήτων, πυρηνική προσωμείωση και επικοινωνία και δημόσιες σχέσεις. Για την ε, εκπαίδευση έχουμε δημιουργήσει ένα πρόγραμμα, νέο πρόγραμμα Master. Ε, είναι για μηχανική για την πυρηνική ασφάλεια. Ε, παίρνει στο τέλος κανείς ένα μάστερ. Είναι ένα συνεχές πρόγραμμα σπουδών, τέσσερα εξάμεινα, δύο χρόνια, πλήρης κύκλος σπουδών και μόλις ξεκινήσαμε τον Οκτώβριο φέτος. Τώρα, το περιεχόμενο των μαθημάτων, ε, ο κύκλος ε, των πυρηνικών ε, καυσίμων, η λειτουργία και η ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων, πυρηνική φυσική και πυρηνική χημεία, τεχνολογία για την επεξεργασία των αποβλήτων και τη διάθεσή τους, προσωμείωση, έχουμε υπολογισμό με υπολογιστές υψηλής επίδοσης, ανάλυση ασφάλειας, διαχείριση των ενεργών αποβλήτων και διάθεση και ο στόχος είναι να εκπαιδεύσουμε πολύ ψηλά καταρτισμένους ειδικού για όλο τον κύκλο ζωής του πυρηνικού καυσίμου. Να αναφέρω ότι ε, στην, το 2009 είχαμε αποφασίσει ότι πριν το Άχεν, Είχαμε μάλλον αποφασίσει πριν το 2005 ότι δεν θα, υπήρχε καθόλου, δεν υπήρχαν καθόλου πυρηνικά στην βόρεια Ρινανία Βεσφαλία, αλλά μετά το 2005 αλλάξαμε πολιτική. Πάμε τώρα στη μεταστοιχείωση. Καταρχάς, γιατί πρέπει να προβούμε σε μεταστοιχείωση και τι είναι η μεταστοιχείωση. Αν κοιτάξουμε ένα ε, μη ακτινοβολημένο καύσιμο, ένα τόνο, ας πούμε, χίλια κιλά, Ας πούμε, έχουμε το τμήμα του ουρανίου, αν υπάρξει εμπλουτισμός σε 33 βαθμούς, τότε έχουμε 33 κιλά α, ουράνιο 235 στην αρχή. Έτσι. Και μετά από τρία χρόνια στον αντιδραστήρα έχουμε 8 κιλά ε, τέτοιου ουρανίου που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί, που δεν έχουν ακτινοβοληθεί για την παραγωγή ενέργειας. Επιπλέον, έχουμε ως αποτέλεσμα της ε, διαδικασίας χάσης, έχουμε τα προϊόντα χάσης, έχουμε το πλουτόνιο, ουράνιο 236 ε, και τους ε, λάσονες ακτινίδες όπως λέμε, νεπτούνιο, αμερίκιο και κούριο. Το πλουτόνιο και τα τρία τελευταία ραδιονουκλεΐδια έχουν μακρά διάρκεια ζωής. Και αυτά είναι τα στοιχεία που είναι υπεύθυνα για το πρόβλημα ε, που μας, θα μας απασχολήσει στο μέλλον για εκατομμύρια χρόνια σε ό,τι αφορά την τελική ε, διάθεση. Αν, θα μπορούσα, αν μπορούσαμε να καταστρέψουμε αυτά τα ραδιονουκλεΐδια, τότε θα μπορούσαμε να μειώσουμε τις προϋποθέσεις ασφάλειας για τα σημεία εναπόθεσης μακροχρόνια. Λοιπόν, εδώ τώρα βλέπουμε ε, σε ένα, ε, για μια χρονική διάρκεια 100.000 χρόνων τη ραδιοτοξικότητα διαφόρων χημικών στοιχείων. Αυτό που βλέπουμε, ε, βλέπουμε αριστε, δεξιά συγγνώμη, είναι ότι τρία από αυτά τα στοιχεία που είναι υπεύθυνα για την μακρά ραδιοτοξικότητα, πλουτόνιο, αμερίκιο και κούριο, είναι αυτά τα τρία λοιπόν. Αν μπορούσαμε να καταστρέψουμε αυτούς τους, αυτά τα ραδιονουκλεΐδια, τότε θα μιλούσαμε για ασφάλεια μετά από τα χίλια χρόνια σε σχέση με το μη ακτινοβολημένο ουράνιο. Τώρα, ποιο είναι το πολιτικό σκηνικό στη Γερμανία ε, και τι, τι συζητάμε σε σχέση με την τελική διάθεση. Το θέμα η λύση η ε, ραδιενέργειας. Ε, έχει επιληθεί αυτό, ε, δημιουργώντας το κόντρατ που είναι ένα τελικό σημείο διάθεσης που πήρε άδεια το 2002 για τη λειτουργία του και τώρα είναι υπό κατασκευή. Θα αρχίσει να λειτουργεί κάποια στιγμή μεταξύ του 2015 και 2019. Τώρα για τα πολύ ραδιενεργά απόλυτα, απόβλητα, στη Γερμανία το τελικό σημείο εναπόθεσης το αναζητούμε ακόμα. Και η όλη διαδικασία θα μπορούσε να ξεκινήσει το νωρίτερο το 2035, εάν μπορούμε να αποδείξουμε την καταλληλότητα του χώρου. Φυσικά αυτό έχει τεράστια πολιτική σημασία στη Γερμανία Οπότε θα φανταστείτε ότι θα έχουμε συζητήσεις και στο μέλλον. Γιατί θα πρέπει να αναζητήσουμε ενδεχομένως και άλλες εναλλακτικέ λύσεις σημείων αναπόθεσης. Προς το παρόν δεν έχουμε όμως τελική, τελικό σημείο διάθεσης για τα πολύ διενεργά απόβλητα. Τώρα, αν συγκρίνουμε τις ε, διαφορετικές στρατηγικές διαχείρισης των αποβλήτων. Βλέπετε σε αυτό το γράφημα στα δεξιά έχουμε το χρόνο μέχρι 10 εκατομμύρια χρόνια και τον πιθανό κίνδυνο στον αριστερό άξονα. Εάν δεν κάνουμε τα τίποτα, αν απλώς ε, διαθέσουμε οριστικά τα ακτινοβολημένα καύσιμα ε, βλέπετε, έχουμε την δεξιά, την, την κόκκινη γραμμή. Αν κάνουμε επανεπεξεργασία του ουρανίου και του πλουτονίου, θα φτάναμε στην ε, κίτρινη γραμμή. Εάν κάνουμε ε, διαχωρισμό, που είναι επανεπεξεργασία και μετά μεταστοιχείωση για την καταστροφή αυτών των ραδιονουκλεϊδίων που σας μίλησα, τότε καταλήγουμε στην πλέγραμμη. Συνολικά λοιπόν, θα φτάσουμε σε μείωση ενός παράγοντα 1 προς 10 σε σχέση. Δηλαδή, κόκκινη με μπλε γραμμή έχουν μια διαφορά 1 προς 10. Τώρα, ποια είναι η αρχή της μεταστοιχείωσης. Πώς καταστρέφουμε τα μακρόβια ε, σωματίδια. Εδώ βλέπουμε το παράδειγμα ε, του πλουτονίου 239 χρειαζόμαστε νετρόνια για να τα καταστρέψουμε αυτά. Αλλά αυτά τα νετρόνια για να τα παράγουμε χρειαζόμαστε καταρχάς πρωτόνια από πυρήνε και θα πρέπει να τα επιταχύνουμε αυτά πρωτόνια και συνεχεία να τα θερμάνουμε ε, με ένα, να έχουμε ένα στόχο ε, διαχωρισμού που θα δημιουργήσουμε από ένα πρωτόνιο και 20 νετρόνια. Και αυτά τα νετρόνια χρησιμοποιούνται για να υπάρξει σχάση των τεσσάρων αυτών ραδιονουκλεϊδίων για τα οποία σας μίλησα προηγουμένως και θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε κάποια προϊόντα σχάσης τα οποία έχουν μικρότερο χρόνο ζωής ή δεν ε, είναι καθόλου ραδιενεργά. Τώρα, ερευνούμε την μεταστοιχείωση για ένα μηχανισμό που ψύχεται με αέριο, διαφορετικό από αυτό που κάνουν στη Γαλλία στο Βέλγιο. Θα το εξηγήσω αυτό σε λίγο. Έχουμε διάφορους εταίρους ε, στα προγράμματα. Είναι το Ινστιτούτο μου στο Άχεν, ας πούμε, είναι αυτό. Έχουμε ένα αριθμητικό κέντρο στο Γιούλιχ. η Ζήμεν συμμετέχει. Έχουμε το, το Ινστιτούτο Φραγκφούρτης ε, προηγμένων επιστημών. Αναπτύσσουμε ένα δημιουργούμε ένα πείραμα μεταστοιχείωσης ε, που λειτουργεί με ε, επιταχυντή, ε, που λειτουργεί με υποκρίσιμο αέριο. Τι σημαίνει υποκρίσιμο. Χρειαζόμαστε δηλαδή έναν επιταχυντή, ούτω ώστε το μηχάνημα να γίνει κρίσιμο. Αν κλείσουμε τον επιταχυντή, τότε η διαδικασία θα σταματήσει πάρα αυτά. Οι στόχοι θα πρέπει να είμαστε συμβατοί με μια πολιτική α, βαθμιαίας εξάλληψης. Ε, ψάχνουμε υποκρίσιμα συστήματα και κάνουμε και μια μελέτη σκοπιμότητας. Ξεκινήσαμε τη μελέτη αυτή τον Οκτώβριο 2008 και θα δημοσιεύσουμε τα, τα αποτελέσματα το Φεβρουάριο του 2011 το Ινστιτούτο μου, μαζί με τους διάφορους εταίρους, μέσα σε αυτό το κρίσιμο, ε, σε αυτό το λίγο χρονικό διάστημα κάνει αυτά τα πράγματα, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες. Το βασικό θέμα είναι φυσικά τα πυρηνικά καύσιμα. Ε, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα επιταχυντή επαρκή για όλο το σύστημα, να αναζητήσουμε την πηγή των νετρονίων και τι μορφή θα έχει ο στόχος ε, διαχωρισμού. Ε, χρησιμοποιούμε τη μετρονική και τη θερμική υδραυλική που είναι χρήσιμη, που είναι απαραίτητη μάλλον για τον ε, αντιδραστήρα που ψύχεται με το υποκρίσιμο αέριο και τα ωφέλη από αυτή την τελική διάθεση των πολυραδινεργών αποβλήτων. πρέπει να δούμε Ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα της μεταστοιχίωσης λοιπόν και αν έχει όφελος, ας πούμε, αν μας δίνει όφελος για την τελική διάθεση των αποβλήτων. Λοιπόν, τώρα, γύρω από το στόχο διαχωρισμού, τα στοιχεία των πυρηνικών καυσίμων βρίσκονται και φυσικά έχουμε και ένα μηχανισμό θωράκισης. Τώρα, ποια είναι τα διάφορα συστήματα και τα διεθνή προγράμματα. Έχουμε καταρχήν τέσσερι, διαφορετικές προσεγγίσεις. Καταρχάς, έχουμε τη γαλλική προσέγγιση, Astrid, έναν γρήγορο ε, αντιδραστήρα που ψύχεται με νάτριο. Το αλέγκρο, επίσης γρήγορο αντιδραστήρα, από την Τσεχική Δημοκρατία, την Τσεχία ε, και τη Σλοβακία. Μετά Έχουμε γρήγορο ε, αντιδραστήρα που ψύχεται, υποκρίσιμο, που ψύχεται με ε, μόλυβδο και βυσμούθιο. Ε, λειτουργεί με τρόπο ADS, ε, κρίσιμο ή υποκρίσιμο σύστημα. Και εμείς ε, προτείνουμε ένα άλλο σύστημα με εστίαση στην μεταστοιχείωση που ψύχεται με αέριο. Ο αντιδραστήρας δηλαδή ψύχεται με αέριο. Τώρα, αν συγκρίνουμε αυτά τα δύο ε, υποκρίσιμα συστήματα, αγκάτε μοίρα, ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια είναι τα μειονεκτήματα εκάστου. Καταρχάς, τα πλεονεκτήματα του μοίρα ε, με βυσμούθιο ε, και, ή μόλιβδο είναι ε, μεγαλύτερη δυνατότητα το ψυκτικό να αντέξει υψηλές θερμοκρασίες και λιγότερο λειτουργικό μεγαλύτερη λειτουργική δυνατότητα. Τα μειονεκτήματα, διάβρωση, ε, ε, Συγγνώμη, μάλλον τα πλεονεκτήματα του αγκάθε είναι ε, απλουστευμένος χειρισμός του στοιχείου του καυσίμου, απλούστερη από ραδιενεργοποίηση, ε, πλεονεκτήματα στην διαδικασία διών, αν κοιτάξουμε το σύστημα με μόλιδο, όλα τα νετρόνια ε, δημιουργούνται μέσα σε 50 ε, εκατοστά. Ενώ στο άλλο σύστημα, λόγω της δυνατότητα να έχουμε ένα πιο συγκεκριμένο στόχο, μπορούμε να κάψουμε, να κάψουμε τα μακρόβια σωματίδια Τώρα, το επόμενο βήμα. Ε, μετά το... τη συζήτηση Βέλγων και Γερμανών, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων, διαβούλευση, διαδικασίες διαβούλευσης για να αναπτύξουμε το πρόγραμμα Αγκάτε. Συμπεράσματα. Ε, ο διαχωρισμός και η μεταστοιχείωση, ε, αν γίνουν, ε, μπορούν να οδηγήσουν στη μείωση της ραδιοτοξικότητας των πολύ ανεργών αποβλήτων. το υποκρίσιμο αυτό σύστημα με επιταχυντή είναι κατάλληλο για τη μείωση αυτών, της ραδιενέργειας των πολύ ραδιενεργών αποβλήτων. Επίσης, η μελέτη σκοπιμότητας θα αποδείξει τις, θα δείξει μάλλον ποιε είναι οι τεχνικέ προδιαγραφέ αυτού του συστήματο. Επίση, θα χρειαστούμε άλλα 20 χρόνια για να αποδείξουμε ότι έρευνα και ότι υπάρχει τεχνική δυνατότητα να φτιάξουμε αυτό το μηχανισμό μεταστοιχείωσης. Αυτά και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Äh, Θέλω να ευχαριστήσω για τις ενδιαφέρουσες επιπρόσθετες πληροφορίες και τώρα θα ολοκληρώσουμε τον πρώτο γύρο με ορισμένα σχόλια του δόκτορα Άπελ και του δίνω το λόγο σχετικά με την διάθεση τον, ε, ε, σε βαθιά γεωλογικά υποστρώματα. Μου ζητήθηκε να μιλήσω για την ε, επιλογή των σημείων εναποθέσεως από την πλευρά του κοινού, διότι εδώ πρόκειται για την ουσία του σχεδίου της οδηγίας και θα αναφερθώ σε τρία σημεία και μετά στη λεπτομέρεια. Καταρχήν τις υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας που πρέπει να υπάρχουν ή στην διαφάνεια των διαδικασιών λήψεως αποφάσεως και της ε, συμμετοχής ε, των, ε, του κοινού στην λήψη αποφάσεων αντιλαμβάνεστε ότι εδώ πέραν των θεμάτων ασφαλείας προκύπτουν θέματα κοινωνικά που είναι πολύ σημαντικά και εδώ θα αναφερθώ ουσιαστικά σε επιγραμματικά στα σημεία που εμφανίζονται στο γράφημα και θα το, τα σχολιάσω διότι υπάρχει διαφορετική ε, διαμόρφωση στα διάφορα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρειάζονται διαφορετικές λύσεις οι οποίες πρέπει να προσαρμοστούν ε, και στο πολιτικό και στο γεωλογικό υπόβαθρο πρέπει δηλαδή να είναι προσαρμοσμένες οι λύσεις στο γενικό πλαίσιο. Καταρχήν θα ήθελα να σας υπενθυμίσω σε γενικές γραμμές γιατί σήμερα ε, ζητούμε να υπάρχει σημείο εναπόθεσης ε, βαθιά στο υπέδαφος ε, διότι καταρχήν η απόσταση μεταξύ των αποβλήτων και της βιοσφαίρας λόγω της γεωλογίας είναι η σωστή λύση επίσης πρέπει τα ραδιενεργά στοιχεία να αποκλειστούν και ε, να μην μεταφερθούν τα, οι αρνητικές τους επιδράσεις μέσω του νερού ή αερίων ε, δεν πρέπει να χρειάζονται συνεχή παρακολούθηση ε, και διόρθωση και επίσης αυτή η παθητική κατάσταση πρέπει να συγκριθεί με την, ε, ε, με το χρονικό περιθώριο το οποίο πρέπει να συνδυάζεται που πρέπει να είναι ε, βραχή και τέλος να υπάρχει ένα συγκεκριμένο σημείο το οποίο έχει εντοπιστεί και το οποίο μπορεί κανείς να αποδείξει τη λειτουργικότητα και την, και την ασφάλεια. Παλιά λέγαμε ότι ήταν και ε, θέμα κόστους, πράγμα το οποίο αυτή τη στιγμή είναι πιο επουσιώδη σημασίας. Αλλά υπήρξε ε, μία συγκεκριμένη συγκέντρωση σε αυτά τα σημεία εναπόθεσης ε, και διαπιστώσαμε ότι ε, ε, υπάρχουν όχι μόνο προσόντα αλλά και μειονεκτήματα λόγω της μακροπρόθεσμης παρακολούθησης που δεν είναι δυνατή και διότι ξεκινάμε για χρόνο αποδομήσεως ο οποίος είναι ενός εκατομμυρίου ετών και αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι δυνατόν να περιοριστεί όπως μας ελέγχθη. Επιπλέον έτσι δεν μπορεί να εγγυηθεί κανείς ότι θα υπάρχει μακροπρόθεσμη παρακολούθηση και πρέπει να υπάρξει χιστρέβλωση μέσα στο χρόνο. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει συντήρηση και επιδιόρθωση και επιπλέον δεν είναι μία βιώσιμη λύση και μακροπρόθεσμα. Ε, επίσης λόγω των χρονικών παραμέτρων και του περιπλόκου χαρακτήρα της διεργασίας δεν είναι δυνατό να βασίσει κανείς τις αποφάσεις σε αποδεδειγμένες επιστημονικές διαπιστώσεις διότι υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία δεν είναι πλήρως κατανοητά. Υπάρχει ακόμη αρκετή ασφάλεια την οποία βέβαια πρέπει ανασφάλεια την οποία πρέπει να μειώσουμε. Όσο αναφορά την επιλογή λανθασμένου σημείου δεν μπορεί κανείς να την διορθώσει αφού αποκλειστούν τα αντικείμενα αυτά στο σημείο εναπόθεσης. Γι' αυτό και προσπαθούμε ε, σοβαρά να μειώσουμε τις ασάφειες επιστημονικά και με έρευνες κατά τρόπον ώστε να έχουμε ένα ισχυρό σύστημα το οποίο θα θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις προσμονές μας. Ε, όλα αυτά δεν έχουν αντιμετωπιστεί θετικά από όλους και στη δημόσια γνώμη ε, δημιουργήθηκαν ε, από την αρχή αμφιβολίες, ζητήθηκε να βρεθούν άλλες λύσεις, ιδίως όταν επρόκειτο για σημεία αναπόθεση κοντά στον τόπο κατοικίας των ενδιαφερομένων και ζητήθηκαν τέτοιες άλλες λύσεις ιδίω με ένα σύστημα το οποίο θα επιτρέπει την εναπόθεση αλλά και την ε, ε, δυνατότητα απομακρύνσεως και πάλι από αυτό το σημείο. Οπότε ε, θα ψάχνουμε να βρούμε με ποιο τρόπο θα μπορούσε κανείς τα απόβλητα αυτά να τα απομακρύνει από το αρχικό σημείο εναποθέσεως ε, με ασφάλεια. Ε, η συζήτηση μεταξύ τεχνικών και εμπειρογνωμόνων έχει αναπτυχθεί μαζί με το κοινό και διαπιστώθηκε ότι ε, η τελική εναπόθεση σωστά έχει ε, αποφασιστεί και ε, το τέλος της δεκαετίας του 70 και στις αρχές του 80 προγραμματίστηκαν εθνικά τέτοια σημεία εναπόθεσης ε, τα οποία βέβαια οδήγησαν σε αντιδράσεις μετά σε καθυστερήσεις και σε διακοπή των προγραμμάτων σε πολλές περιπτώσεις. Επίσης αυτό οδήγησε στο ότι οι υπεύθυνε αρχές ασχολήθηκαν με τις ανησυχίες των ενδιαφερομένων, χρειάστηκε να τους απαντήσουν και έκτοτε υπησήλθε στη συζήτηση και το θέμα των επιφυλάξεων των ενδιαφερομένων ομάδων ή του πληθυσμού που κατοικεί στην ε, περιοχή και η συζήτηση έχει ε, ε, οξυνθεί πολύ περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Στη δεκαετία του 80 συνεχίστηκε αυτή η κατάσταση και έκτοτε η ε, αντιπαράθεση μεταξύ των κοινωνικών στοιχείων και των επιστημονικών οδήγησε σε οξυμένη συζήτηση. Τώρα πια δεν υπάρχει συζήτηση ε, διότι τώρα πλέον δεν υπάρχει ποτέ συζήτηση χωρίς να προσθέτει κανείς τους όρους ε, διαφάνεια, ισότητα α, ε, δίκαιο και δυνατότητα ε, μετατοπίσεως αυτών των προϊόντων, των αποβλήτων. Ε, έχουν υπάρξει συμφωνίες σε ορισμένα σημεία και από το τέλος της δεκαετίας του 90 και το 2000 όπως ακούσατε έχουν καταρτιστεί διάφοροι οργανισμοί οι οποίοι ασχολούνται συγκεκριμένα με αυτά τα θέματα και θα μπορούσα εδώ να αναφερθώ και στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, το πρόγραμμα COVAM που διεξήχθη 2000 έως το 2009 σε τρεις φάσεις. COVAM σημαίνει Community Waste Management όπου σαφώς αναφέρεται ότι πρέπει κανείς να ασχοληθεί και με τις ανησυχίες του κοινού, του πληθυσμού που διαβεί στην περιοχή και ε, στην αρχική φάση όταν συζητά κανείς τη στρατηγική θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι της περιοχής να μην αισθάνονται ότι εμπλέκονται στο θέμα και στη συνέχεια συγκεντρώνονται, οργανώνονται και όταν πλησιάζει η απόφαση τότε αντι αντιλαμβάνονται ότι πρόκειται να υπάρξει ένα τέτοιο σημείο αναπόθεση κοντά στις κατοικίες τους και αντιδρούν. Βεβαίως ιστορικά βλέπουμε ότι φτάνει κανείς σε ένα σημείο της συζήτησης και το έθιξα προηγουμένως, δηλαδή βλέπουμε πώς αυτή τη στιγμή αντιδρύουν αυτές οι ομάδες των κατοίκων. Βλέπουμε από το 2001 όπου το ότι θα υπάρξει τελική εναπόθεση ε, των ραδιενεργών βλήτων που θεωρείται στην αρχή πολύ επίγουσα και πολύ σημαντική ε, μέχρι 53% των ενδιαφερομένων αλλά όταν τους ρωτούσε κανείς τι θα γίνει με το τελικό σημείο εναπόθεσης θέλεις να είναι στην περιοχή σου οπότε 80% απαντούσαν όχι όχι όχι κοντά σε μένα οπότε από τη μία πλευρά πρέπει να γίνει αποδεκτή η ανάγκη αλλά από την άλλη μεριά διαπιστώνουμε ότι υπάρχει αντίφαση διότι δεν θέλουν αυτό το σημείο εναπόθεσης να είναι κοντά στι κατοικίε τους και εκεί τίθεται ένα θέμα το οποίο πρέπει κανείς να αντιμετωπίσει. Ακόμη και σήμερα, στο 2010 δηλαδή, διαπιστώνουμε ότι στα αποτελέσματα της διαβουλεύσεως με το κοινό για την επεξεργασία της οδηγίας υπάρχουν ορισμένες προτιμήσεις. Πρέπει να προστατευτούν οι επόμενες γενιές από τις επιδράσεις της ραδιενεργίας, να υπάρχει ε, διαφάνεια, το λέει το 64%. Ε, να υπάρχει ανεξαρτησία της ρυθμιστικής αρχής 64% αλλά ελάχιστοι θέλουν βιολογική τελική εναπόθεση. Δηλαδή η βιολογική εναπόθεση συναντά αντίσταση από τους ενδιαφερόμενους, από την κοινή γνώμη γενικώ, από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις οι οποίες τοποθετούνται και ε, αποφασίζουν ε, βάσει των αρχών τους και βλέπετε εδώ τα αποτελέσματα μίας μελέτης σχετικά με το πρόγραμμα COVAM και ε, εδώ θα ήθελα να αναφερθώ μόνο σε συγκεκριμένα σημεία στο D, B comprehensive δηλαδή να σκεφτείτε σφαιρικά και τεχνικά και κοινωνικά να συμμετάσχουν πέρα των τεχνικών και όλοι όσοι ενδιαφέρονται για τη διαδικασία. Ε, επίσης να υπάρχει μία πλήρης συμμετοχή και να επηρεάζουν, να μπορούν να επηρεάσουν οι συμμετέχοντες. Ε, εδώ είναι το ευχολόγιο των ενδιαφερομένων που ε, έχουν συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία και ο κύριος Ριώτο ανέφερε ε, την δυνατότητα βέτο των ορισμένων Πού καταλήγουμε λοιπόν για τη διαδικασία επιλογής ενός σημείου εναποθέσεως σήμερα δεν είναι απαραίτητο στη συζήτηση για την τελική εναπόθεση να αποδείξει κανείς ότι το, η στρατηγική αυτή την οποία χρησιμοποιούμε είναι η πλέον ασφαλής. Δηλαδή πρέπει να είναι η πλέον ασφαλής για την περιοχή στην οποία οργανώνεται η εναπόθεση. Ε, οπότε θα πρέπει οι κάτοικοι και οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν διότι σας είπα ότι στην αρχή είναι δύσκολο να συμμετάσχουν όλοι γιατί οι ε, ε, κάτοικοι της περιοχής αισθάνονται ότι εμπλέκονται πρέπει να αναγνωρίσει κανείς ότι οι περιοχές στην οποία γίνεται η τελική ε, εναπόθεση πρέπει να ανταμυφθούν για την προσφορά τους και πέραν της ε, ε, ε, αμοιβή θα πρέπει να υπάρχει και μία γενικότερη περιφερειακή αντιμετώπιση θετική της προσφοράς. Συνοψίζοντας, όσον αφορά τα αντικρουόμενα αυτά συμφέροντα και τις απόψεις τα οποία απεικόνισα, όπου επιζητείται μια πιο ασφαλής λύση πρέπει να δούμε ποιες δέχεται να είναι οι επιπτώσεις. Δηλαδή πόσο μπορεί κανείς να συνδυάσει τις τεχνικές και τις μη τεχνικές απόψεις ε, είναι κάτι πολύ δύσκολο μεθοδολογικά και στο μέλλον θα είναι δύσκολο να συνδυαστούν αυτά τα στοιχεία διότι δεν υπάρχει προστιθέμενη αξία στις απόψεις αυτές οι οποίες πρέπει να ληφθούν υπόψη για την επιλογή ενός σημείου εναπόθεσης δεν μπορούμε πούμε ότι υπάρχει μία επιπρόσθετη αξία, μία προστιθέμενη αξία για την επιλογή του σημείου. Και μάλιστα δεν προχωράμε με αυτά τα κριτήρια διότι δεν θα μπορούμε να καταλήξουμε σε καμία απόφαση. Ο στόχος είναι αυτός ο οποίος εκφράζεται στην αρχή safety first, πρωτεύει η ασφάλεια. Και μόνο αν εφαρμόσουμε αυτή την αρχή ή θα μπορέσουμε να πείσουμε ε, τους κατοίκους με σωστά επιχειρήματα περί της ασφαλείας ότι ακόμη και αν δεν τους αρέσει θα πρέπει να δεχθούν ότι θα υπάρχει ένα σημείο εναπόθεσης κοντά στις κατοικίες τους. Ίσως θα είναι πιο εύκολο να πιστούν όταν η διαδικασία αυτή αποδεικνύεται μεθοδολογικά όπως προανέφερα η αρχή αυτή του safety first σημαίνει ότι υπάρχει μία προτεραιότητα της ασφαλείας, δηλαδή των τεχνικών απόψεων ε, έναντι των μη τεχνικών. Και μόνο όταν εξαλειφθούν οι τεχνικοί κίνδυνοι μπορεί κανείς να περιλάβει ε, άλλες απόψεις σε αυτή τη διαδικασία. Και με <clears throat> αυτά τα τελικά σχόλια ε, κλείνω την παρουσίασή μου. Ελπίζω ότι ε, διευκρίνησα το θέμα μου και δεν σας άφησα σε αμφιβολία διότι ε, τα τρία τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί διαδικασίες ε, και χρησιμοποιούνται στα συμμετέχοντα κράτη-μέλη όχι μόνο για να πιστούν οι άνθρωποι αλλά για να χρησιμοποιηθούν διαδικασίες λήψεως αποφάσεων που να προσαρμόζονται στις ε, γενικές διαδικασίες που επιτρέπουν να καταλήξουμε σε μία ασφαλή και χρήσιμη λύση. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ähm, ευχαριστώ. Έτσι Ολοκληρώσαμε το, την πρώτη ενότητα πληροφοριών και τώρα συνάδελφοι έχετε τη δυνατότητα να κάνετε ερωτήσεις για να ζητήσετε επιπρόσθετες παρατηρήσεις. Ο κύριος Τσουκαλάς είναι ο πρώτος και θα παρακαλούσα να θέτετε ως το δυνατόν πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις για να έχετε και συγκεκριμένες απαντήσεις. Ο κύριος Τσουκαλάς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τους ε, κυρίους ε, του πάνελ. Μας έδωσαν πολύτιμες πληροφορίες ε, που σχετίζονται και με την δουλειά μας εδώ. Θα ήθελα να κάνω την εξή γενική ερώτηση, κύριε Πρόεδρε, δοθέντως ότι ακόμα και στις πιο αισιόδεξε εκδοχές, αν παραδείγματι, όπως είπε ο καθηγητής κύριος Τόμαουτς μπορούσαμε να εξαφανίσουμε τα ακτινίδια, θα μιλούσαμε για ασφάλειες ε, της, της τάξεως των χιλίων ετών, αλλιώς θα μιλούσαμε για ασφάλειες της τάξεως του ενός εκατομμυρίου ετών. Η συζήτηση οξυμένη που ανέφερε ο κύριος Άπελ και η οποία πράγματι είναι μία ανάμιξη επιστήμης, προκαταλήψεων και ανησυχιών, είναι μια συζήτηση που θα εξακολουθήσει να μας ε, ταλαιπωρεί δοθέντως το ότι σύμφωνα με όλα τα δεδομένα φαίνεται ότι αν εξακολουθήσουμε να έχουμε τον ίδιο τύπο ανάπτυξης με τους ίδιους ρυθμούς ανάπτυξης με το 2025 να βλέπει την ανθρωπότητα με 8 δισεκατομμύρια κατοίκους με ραγδαία ανάπτυξη των χωρών της Ασίας και του Ειρηνικού τότε είναι προφανές ότι αν διατηρηθεί η ανακεφαλή κιλοβατόρα, τότε οι ενεργειακές ανάγκες της ανθρωπότητος στο πρώιμο στάδιο της ανάπτυξης των εναλλακτικών μορφών ενέργειας φαίνεται να είναι απαραίτητο να ακουμπήσει στην πυρηνική ενέργεια. Στην πυρηνική ενέργεια την οποία είναι κάτοικοι όλων των κρατών με μεγάλη δυσπιστία βλέπουν και μεγάλη ε, επιφυλακτικότητα αντιμετωπίζουν. Η πρόσφατη επίθεση του Bill Gates εναντίον της αποδόσεως των εναλλακτικών μορφών ενέργειας όπως αυτές είναι σήμερα, δηλαδή στο επίπεδο του 10 με 12% και η ταυτόχρονη παρένεσή του να επιδοθούν, να δοθούν πολλά χρήματα για την έρευνα, για την ε, ανακάλυψη νέων τεχνολογιών αναλλακτικών μορφών διαμορφώνει τελικά την ερώτησή μου, την οποία απευθύνω σε εσά, αν μπορείτε να την απαντήσετε, κατά πόσο θεωρείτε ότι η πυρηνική ενέργεια, η χρήση της πυρηνικής ενέργειας, είναι ένα πράγμα το οποίο, επαναλαμβάνω, με τον ίδιο τύπο ανάπτυξης και τον ίδιο ρυθμό ανάπτυξης, τελικά η ανθρωπότητα θα πρέπει να ακουμπήσει αν λάβει κανείς υπόψη του ότι σε διάφορες χώρες της Ευρώπης αλλά και στη Βόρεια Αμερική η ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας έχει πάρει φόρα πάλι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Χάρμς έχει το λόγο. Έχω μία ερώτηση στον κύριο Τομάουσκε ή μάλλον δύο ερωτήσεις και εδώ αναφέρομαι σε ποιο στάδιο ανάπτυξης βρίσκονται αυτοί οι αντιδραστίες ε, για την partition ή την transmutation, ε, δηλαδή ε, για τον διαχωρισμό ή την μεταστοιχείωση πόσο δαπανηρή είναι αυτά τα προγράμματα, ποιος τα χρηματοδοτεί και ε, πού μπορεί κανείς ε, να θεωρήσει ότι η μεταστοιχείωση είναι ε, ένα μέρος της στρατηγικής εναπόθεσης. Επίσης προς τους κυρίους Ριώτε και Άπελ. Ε, όσον αφορά την, ε, ε, την ε, διατύπωση που περιέχει η οδηγία του Επιτρόπου Ότιγκερ, δηλαδή ότι υπάρχουν πολλές χώρες όπου υπάρχει συνένεση να υπάρξουν βαθιά γεωλογικά σημεία εναπόθεσης και θα αποτελέσουν την καλύτερη λύση. Δηλαδή ποια είναι η ποιότητα αυτής της συνενέσεως, ποιος συμφώνησε με ποιον. Κύριε Ριώτε, αυτό περιέχει και αυτό που είπατε εσείς, ε, δηλαδή ε, μία κοινωνική αποδοχή ενός τέτοιου προγράμματος βαθιάς ε, ταφής γεωλογικής ε, των αποβλήτων επίσης ε, κύριε Άπελ και κύριε Ριώτε για ποιες χώρες ε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λύση αυτή των, της βαθιάς ταφής γεωλογικά των πολύ ραδιενεργών αποβλήτων και πού υπάρχει συμφωνία που έχουν διακοπεί ε, αυτά τα προγράμματα και επίσης θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται και ε, ε, το θέμα της απομακρύσεως ορισμένων κλειστών αποβλήτων από το χώρο της ΆΣΕ. Πώς αυτά εντάσσονται σε όλο το πρόγραμμα της ταφής και μετά της επιστροφής. Θα ήθελα και εγώ εγώ να κάνω μία ερώτηση προς τον κύριο Τομάους και, ε, γιατί συνδυάζεται με την ερώτηση της κυρίας Χάρμς και θα ήθελα να προχωρήσω περαιτέρω γιατί είναι μία ενδιαφέρουσα προσθήκη. Κύριε Τομάους και χρονικά αυτό το σενάριο εάν συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε αυτό το πρόγραμμα πότε θα επιτύχουμε τι, ποιον στόχο γιατί αυτό είναι το επόμενο. Επίσης ο συνάδελφος Κούτσικ. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που οργανώσατε αυτή την ακρόαση. Νομίζω ότι είναι πραγματικά έρχεται την κατάλληλη στιγμή. Θα ήθελα να ρωτήσω καταρχήν τον κύριο Τομάουσκε Τα σχέδια στα οποία αναφερθήκατε αποτελούν τμήμα του καταλόγου ε, που γνωρίζουμε. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα λοιπόν και πότε νομίζετε ότι θα έχουμε τα πρώτα απτά αποτελέσματα. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναφερθεί πάρα πολύ στο γεγονός ότι αυτό ο κατάλογος ε, σχεδίων θα πρέπει να προχωρήσει και δεν αρκεί να εντάσσουμε συνέχεια ε, projects σε αυτόν τον κατάλογο. Πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή θα, θα πρέπει να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση που θα είναι η εφαρμογή. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε χρονικά πότε το για πότε προβλέπετε. Μια γενικότερη ερώτηση. Μιλάμε για διαχείριση πολύ ραδιενεργών αποβλήτων. Ένα από τα βασικά ερωτήματα λοιπόν είναι το τι θα γίνει. Θα το κάνουμε μονομένα τα κράτη-μέλη ή μπορούμε να δώσουμε μια λύση η οποία θα είναι κοινή όπου θα έχουμε κοινή διαχείριση ή διάθεση αποβλήτων από σύνολο κρατών μελών που χρησιμοποιούν πυρηνική ενέργεια. Δηλαδή, ε, κατά τη γνώμη σας, πόσους χώρους εναπόθεσης θα έπρεπε να έχουμε ε, στην Ευρώπη. Ξέρετε πως η ενέργεια αποφασίζεται από τα κράτη-μέλη. Αν λοιπόν είναι λίγα τα κράτη-μέλη τα οποία χρησιμοποιούν πυρηνική ενέργεια, θα έπρεπε ενδεχομένω να αλλάξουμε τη διαδικασία λήψη απόφαση. Ρωτώ λοιπόν του ομιλητέ, πολύ καλά κάνετε σε περιφερειακό, εθνικό, τοπικό επίπεδο κάποιε έρευνε και μελέτε. Όταν όμω υπάρχει μετακίνηση και μεταφορά μεταξύ κρατών μελών, τότε θα πρέπει στη διαδικασία λήψη απόφαση αυτό να λαμβάνεται υπόψη. Γιατί βέβαια εκεί έχουμε και την αντίδραση ε, του κοινού ε, για τα θέματα αυτής της μεταφοράς. Τι πιστεύετε λοιπόν πως θα πρέπει να γίνει. Ευχαριστώ πολύ. Έχω μια πολύ απλή ερώτηση να κάνω και είναι κάτι το οποίο ρώτησε η κυρία Χάρμς προηγουμένως. Δηλαδή, για την ε, έρευνα που κάνετε. Μπορείτε να μου πείτε πότε προβλέπετε να έχετε μια καλή ιδέα για το γενικότερο κόστος αυτής της προσπάθειας, δηλαδή έναν αντιδραστήρα μεταστοιχείωσης με με, που θα χρησιμοποιεί εξαντλημένα πυρηνικά καύσιμα. Γιατί θα ήθελα να κάνω έναν υπολογισμό του κόστους ε, για να ξέρω ποιο θα είναι το οικονομικό βάρος αυτής της ε, πανεπεξεργασίας ε, των πυρηνικών καυσίμων, γιατί βέβαια ε, συνδυάζεται και με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα ακρόαση που μας οργανώσατε. Πιστεύω πως στην Ευρώπη και στην, στον κόσμο γενικότερα αντιμετωπίζουμε μια παράδοξη κατάσταση. Δηλαδή αντιμετωπίζουμε προκλήσεις όπως η αλλαγή του κλίματος, τα κοινωνικά θέματα που αποβραίνουν από αυτήν, την πυρηνική ενέργεια και το θέμα της διάθεσης των πυρηνικών αποβλήτων. Όλοι γνωρίζουν τι πρέπει να γίνει και απαιτούν οι πολίτες από τις κυβερνήσεις και από του πολιτικούς να δώσουν κάποιες λύσεις. Παράλληλα όμως ελπίζουν πως οι λύσεις αυτές δεν θα τους αφορούν άμεσα. Για να δούμε λοιπόν για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας τι μπορούμε να κάνουμε. Αγοράζουμε όλο και μεγαλύτερο εξοπλισμό, υπερθερμαίνουμε τις κατοικίες μας, αφήνουμε τις συσκευές αναμένες, αφήνουμε τα φώτα αναμένα και ζητάμε από τους πολιτικούς παράλληλα να δράσουν. Νομίζω ότι αυτή είναι μια παράδοξη κατάσταση την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε κατάματα. Δηλαδή, θα πρέπει και η ακαδημαϊκή κύκλη και η βιομηχανία και η πολιτική να μιλήσουμε με μεγαλύτερη σοβαρότητα για τα θέματα αυτά. Δεν θα πρέπει να σκεφτόμαστε μόνο το πώς θα τα εκφράσουμε ε, ε, έτσι ώστε να είναι ικανοποιημένο ε, το ευρύ κοινό. Δηλαδή θα πρέπει τα θέματα αυτά να τα παρουσιάσουμε με ένα σαφή τρόπο έτσι να γνωρίζει ο κόσμος ποια είναι τα προβλήματα που τον περιτριγυρίζουν και να δούμε και η λήψη απόφασης για αυτά τα τόσο βασικά θέματα πώς μπορεί να ε, ανοίξει και σε άλλους παίκτε, να δούμε ποια είναι τα πρότυπα που χρειαζόμαστε για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, από ποιες πηγές θα πρέπει να γίνεται αυτή η παραγωγή και να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε και ασφαλή αποξύλωση όλων αυτών των πυρηνικών εγκαταστάσεων και παράλληλα ασφαλή ε, διαχείριση και διάθεση αποβλήτων. Θα ήθελα για τη μεταστοιχείωση να μου δώσετε κάποιες παραπάνω πληροφορίες. Δηλαδή, οι διαδικασίες αυτές εμπορικά πότε θα θεωρούνται βιώσιμες και ποια είναι τα βασικά εμπόδια μέχρι να γίνει αυτό. Δηλαδή, σας λείπουν γνώσεις, σας λείπουν κονδύλια. Κύριε Τομάουσκα, αναφερθήκατε στα 20 χρόνια που χρειάζεστε πριν τα βάλετε σε ισχύ. Νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε κάπως πιο γρήγορα. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τα πυρηνικά απόβλητα σε κρεμότητα για 20 χρόνια ακόμα. Χρειαζόμαστε τότε να επενδύσουμε περισσότερο σε έρευνα, σε πόρους, γιατί ε, πρέπει να δούμε και τη διάσταση του ποιο θα επενδύσει σε αυτή την τεχνολογία. Δεν θα το κάνει ο ιδιωτικό κλάδο. Γιατί βέβαια ξέρετε πω αυτά τα πολύ ραδιενεργά απόβλητα κάπου ε, κάπως πρέπει να διατηθούν. Θα γίνει μέσω κοντελίων των κρατικών ε, προϋπολογισμών. Η ερώτηση που έκανε η συνάδελφος κυρία Χάρμς ε, με οδηγεί στο εξή συμπέρασμα. Η μεταστοιχείωση μας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τα πυρηνικά απόβλητα με τον τρόπο που χειριζόμαστε άλλου είδους απόβλητα. Άρα λοιπόν το θεωρώ σαν έναν τρόπο ανακύκλωσης. Όμως, για τις χώρες που δεν έχουν τις γεωλογικές συνθήκες που θα τους επιτρέψουν να κάνουν ε, γεωλογική εναπόθεση ή ταφή. Περιφερειακές πρωτοβουλίες υπάρχουν. Θυμάμαι πως για τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης πριν από 15 χρόνια είχε γίνει μια προσπάθεια. Και τότε μας είχαν πει πως δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, δηλαδή υπάρχουν τεχνικές δυνατότητες. Όταν, μας ρωτή, όταν ρωτήσαμε όμως, ωραία, και πού θα βρίσκονται αυτοί τη χώρη διάθεσης, έληξε η συζήτηση. Γιατί ε, κανείς δεν το επιθυμούσε. Και ένα σχόλιο περισσότερο και όχι ε, παρατήρηση και όχι ερώτηση. Είπατε πρώτα η ασφάλεια, όχι μόνο για τη διάθεση των αποβλήτων, αλλά και για την λειτουργία των πυρηνικών εργοστασίων. Δεν νομίζετε κι εσείς πως θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη και το θέμα της κοινωνικής αποδοχής, της επιλογής του χώρου που θα εγκατασταθούν αυτές οι μονάδες. Γιατί νομίζω χρειάζεται να δούμε ε, την κοινωνική συνένεση και αποδοχή πριν περάσουμε στην επιλογή. Γιατί έχω την εντύπωση πως σε επίπεδο κοινωνικής ε, αποδοχής οι γνώμες των εμπειρογνωμόνων δεν μετράνε ιδιαίτερα. Also Λοιπόν, τώρα θα, έλεγα να προσπαθήσετε να απαντήσετε και θα ξεκινήσουμε από το τέλος. Πρώτα ο δόκτωρ Άπελ, μετά ο δόκτωρ Λοριότε και ε, για να αφήσουμε στο τέλος τη μεταστοιχίωση για να μην μπερδεύουμε τα πράγματα. καταρχήν θα απαντήσω στην κυρία Χάρμ. Το πρώτο ερώτημά της αναφερόταν στο, ε, στις χώρες όπου υπάρχει συνένεση σχετικά με τα σημεία εναπόθεσης. Αυτό εξαρτάται ε, από το ποιον θα ρωτήσετε. Δηλαδή, γενικά μπορούμε να πούμε ότι ε, η τελική εναπόθεση ή η αλλαγή του σημείου δεν ε, μπορεί να διαπιστωθεί ότι υπάρχει συνένεση ε, ακόμη και αν ε, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν διαμαρτύρονται ή δεν κάνουν διαδηλώσεις δεν σημαίνει ότι συνενούν. Υπάρχουν όμως άνθρωποι οι οποίοι αισθάνονται ότι απειλούνται και ε, υπάρχει ένας, μια μεγάλη διαφορά μεταξύ της συνένεσης για τη στρατηγική και της συνένεσης για τη διαδικασία στην ε, φάση της εφαρμογής. Και εδώ αναφέρομαι ιδίως στα άτομα τα οποία δεν ε, ε, έχουν επαγγελματικές γνώσεις και συμμετέχουν διότι αισθάνονται ότι είναι ένα θέμα που τους θίγει ή συμμετέχουν για άλλους λόγους στη συζήτηση. Θα προσπαθήσω να σας ε, απαντήσω εμέσως, δηλαδή ποιες χώρες είναι οι πιο προχωρημένες. Ε, το βλέπουμε αυτό σε ποια διαδικασία, σε ποια φάση της διαδικασίας ίσως βρίσκονται ορισμένες χώρες. Αλλά δεν θέλω να προχωρήσω έτσι, γιατί στη Γερμανία είμαστε πολύ προχωρημένοι, αλλά είμαστε σε μεγάλη συζήτηση στη Γερμανία αν αυτό το σημείο εναπόθεση θα παραμείνει ή όχι. Άρα το ότι έχει προχωρήσει η συζήτηση δεν λέει πολλά. Αυτό που είναι πιο σημαντικό είναι η ε, διαδικασία με την οποία καταλήξαμε σε αυτό ε, το σημείο, δηλαδή ε, στη λήψη μιας αποφάσεως ή για τη στρατηγική ή στην επιλογή ενός σημείου. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι προχωρημένες αλλά δεν θα τις σχολιάσω γιατί έχουν διαφορετική διαδικασία αλλά νομίζω ότι η Ελβετία για τα πολύ ραδιενεργά απόβλητα είναι η πιο προχωρημένη ε, ότι πρόκειται για μια διεργασία η οποία έγινε το 1980-90 και επειδή δεν υπήρχε επαρκή στήριξη από πλευράς των καντονιών στην ε, ε, Ελβετία που είναι αρμόδια για αυτές τις αποφάσεις οδήγησε οδήγησε τον αρμόδιο υπουργό τότε να οργανώσει ε, μία δημόσια συζήτηση για την, ε, το μέλλον των ραδιενεργών αποβλήτων. Οπότε δεν ε, κατέληξαν σε μία συνενετική λύση. Στη συνέχεια κατήρτισε μια ομάδα επιρρογνωμόνων όπως κάνει κανείς συνήθως σε αυτές τις, περιουσίες, τις περιπτώσεις που είχε σαν ανηλιμένο καθήκον να ερευνήσει την ταφή των, των ραδιενεργών αποβλήτων σε βαθιά γεωγραφικά, γεωλογικά στρώματα. Έγινε ε, λοιπόν ένα, ε, μία μελέτη η οποία περιελήφθη στην νομοθεσία και καταρτίστηκε ένα σημείο στο οποίο έχει ήδη ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της όλης διεργασίας όπου δηλαδή όλοι οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι μπορούν να παρέμβουν, ακόμη και οι γειτονικές χώρες και ε, πιστεύω ότι εκεί σχετικά σύντομα αυτό βέβαια υποπροϋποθέσεις θα μπορέσει να καταλήξει. Ε, στη Σκανδιναβία υπάρχει επίσης μια τέτοια διεργασία στην Σουηδία και στη Φιλανδία που οδηγεί σε αίσιο πέρας και ε, κατά τη γνώμη μου το δικαίωμα βέτο στη Σουηδία όπου υπάρχει ε, αυτή η ε, νομική διομορφία η οποία υπήρχε και στην, και στην Ελβετία αλλά έχει εξαλειφθεί εντωμεταξύ ε, δεν οδήγησε στην ε, Σουηδία τώρα στην άρση όλων των αποφάσεων αλλά ότι ε, πρέπει να υπάρξει μια συγκεκριμένη διαδικασία για την υλοποίηση αυτών των προγραμμάτων. Και όσον αφορά το τρίτο σημείο, εντοπισμός των αποβλήτων ε, και απόσυρσή τους, έχω σημειώσει μεν την, ε, τα στοιχεία της ερώτησης χωρίς να θυμάμαι ακριβώς τι είχατε πει. Τι με ρωτήσατε. Η ερώτησή μου ήταν η εξής αυτή τη στιγμή ε, ε, ε, ποια είναι η διαδικασία ή ο πολιτικός προγραμματισμός για την τελική εναπόθεση πόσο διαμορφώνονται ιδίως αν λάβει κανείς υπόψη τους ότι υπάρχει ένα Υπουργείο στη Γερμανία το οποίο ανέλευε να ερευνήσει πώς πώς θα μπορούσε κανείς να απομακρύνει ε, αυτά τα απόβλητα από το χώρο εναποθέσεως στο ΆΣΕ. Ε, ναι, υπήρξαν σκέψεις επ' αυτού του θέματος και μπορούμε να πούμε τώρα ότι οι νέες προδιαγραφές της ασφαλείας στη Γερμανία αντικατοπτρίζονται και σε αυτά τα μέτρα, δηλαδή ε, πρέπει να υπάρχει δοχεία τα οποία να μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει ε, για 500 χρόνια παραδείγματο χάρη. Οι διάφορες όμως προτάσεις διαφέρουν πάρα πολύ. Στην ε, Ελβετία έχει ε, επιλεγεί ένα συνδυασμός Δηλαδή προσπαθεί κανείς να αποβλέπει σε μία αφαίρεση για ένα χρονικό διάστημα συγκεκριμένο. Όταν η... τελική συζήτηση περί καθαρής εναπόθεσης ε, και σχετικής εύκολης πρόσβασης στα απόβλητα για να μπορέσει κανείς να τα απομακρύνει είναι τεχνικά τόσο δυσκερές ώστε δεν μπορεί να προχωρήσει. Οι στην λοιπόν διαλέξανε την εξίσοδο. Αφενός συμμετέχει το κοινό ε, στη συζήτηση ε, πότε, πότε ε, πότε έχει λήξει το, η προθεσμία για το θέμα της αφαιρήσεως της αφαιρέσεως από το σημείο εναπόθεσης αλλά και πότε μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι λειτουργεί σωστά το σημείο αυτό. Ε, πρέπει δηλαδή να μπορεί κανείς να παρακολουθήσει το σύστημα και να καταλήξει σε συμπεράσματα. Υπάρχει μία πολύ λεπτομερής διαδικασία η οποία δεν έχει προγραμματιστεί πλήρως αλλά προς αυτή την κατεύθυνση ε, κατευθύνονται και στην ε, Σουηδία ε, υπάρχει μία διαφορετική αντιμετώπιση η οποία άπτεται των γεωλογικών συνθήκων και όπως είπε και προηγουμένως ο κύριος Ριώτη ε, σε ορισμένα συστήματα μπορεί κανείς ε, να ε, απομακρύνει τα απόβλητα από το σημείο εναπόθεσης. Άρα παντού μιλάει κανείς για τα ίδια πράγματα, δυνατότητα απομάκρυνσης αλλά και τεχνικά και πολιτικά πρέπει κανείς να αντιμετωπίσει διαφορετικά τα θέματα αυτά, το πώς μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση σε αυτά τα σημεία και να απομακρύνει από εκεί τα απόβλητα. Και επ' αυτού δεν υπάρχει μία ενιαία αντιμετώπιση. Ε, όπως είπε η κυρία, αν όλες οι μικρές χώρες πρέπει από κοινού να λύσουν το θέμα της απομακρύνσεως των πολύ ραδιενεργών αποβλήτων ή θα πρέπει ε, να υπάρξει μία ενιαία λύση. Στο σημείο αυτό και από πλευράς ε, κοινωνικής, ε, κοινωνικής συνένεσης για ε, ένα κοινό αποδεκτό σημείο εναπόθεσης πιστεύω ότι αυτό θα μπορέσει να επιτευχθεί μόνο αν οι ευθύνε αναλαμβάνονται από κοινού και αυτό μπορεί να αποδειχθεί επιστημονικά διότι δεν είναι δυνατόν μία μικρά χώρα η οποία έχει παράγει ε, ηλεκτρική ενέργεια και απόβλητα και δεν έχει δυνατότητα λόγω της φυσικής θέσεώς της να χρειάζεται να αποθέσει τα απόβλητά της κάπου αλλού, σε μια άλλη χώρα. Αυτό τεχνικώς δεν είναι δυνατόν και γι' αυτό πρότεινα τη λύση την οποία ανέφερα προηγουμένως. Επίσης Αναφερθήκατε στη διαμάχη μεταξύ κοινωνικής αποδοχής και τεχνικών προϋποθέσεων και προσπάθησα να αποφύγω τον όρο αποδοχή και να μιλήσω για τεχνικές πτυχές. Δεν έχω μία τεχνική λύση η οποία να μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ενιαία σε όλη την Ευρώπη διότι οι συγκεκριμένες συνθήκες στην Ευρώπη διαφέρουν από τη μια χώρα στην άλλη, αλλά κατά τη γνώμη μου πρέπει να ισχύσει η αρχή safety first. Δηλαδή αυτό πρέπει να προέχει. Δεν ε, μπορούμε να υποχρεώσουμε να, κάποιον να δεχθεί κάτι ή να σιωπήσει. Και βεβαίως πρέπει να ληφθεί υπόψη και η ιδιομορφία της εκάστοτε χώρας. Ο κύριος Ριώτε. Ίσως θα έπρεπε καταρχήν να επανέλθω στα σημεία τα οποία έθιξε ο κύριος Άπελ ε, δηλαδή εάν ε, εξετάσουμε τα θέματα αυτά της συνενέσεως η γενική απάντηση ε, είναι ε, ότι υπάρχει ε, καταρχήν συνένεση στην Σουηδία, εν μέρη στη Γερμανία, βεβαίως στην Ελβετία και στον Καναδά που έχει καταρτήσει ένα νέο πρόγραμμα πριν από τρία-τέσσερα χρόνια και ένα μέρος αυτού του προγράμματος συνεπάγεται και ένα ερωτηματολόγιο προς όλη την καναδική ε, κοινωνία ε, και νομίζουμε ότι ε, πέτυχαν κάτι το οποίο από μακριά μπορεί να θεωρηθεί σαν συνενετική διαδικασία. Ε, ε, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Σουηδία, η Φιλανδία και η Γαλλία επίσης είναι σε καλό δρόμο από πλευράς χρονολογικής και ιδίως όσον αφορά την αξιολόγηση ε, των επιπτώσεων βρέχει πρόθεσμα. Η Σουηδία και η Φιλανδία στην επόμενη δεκαετία θα υπάρξει εφαρμογή του προγράμματος και στη Γαλλία υπάρχει ήδη το νομικό πλαίσιο. Ε, όσον αφορά την ε, επανάκτηση των στοιχείων αυτών ουσιαστικά ε, υπάρχει η απέτηση η οποία καλύπτεται και ε, νομικά σε πολλές χώρες. Πώς αυτό θα επιτευχθεί είναι ακόμη ανοιχτό. Αλλά στη Γαλλία παραδείγματος χάρη υπάρχει η απέτηση επανακτήσεως εις την νομοθεσία του τελικού σημείου εναπόθεσης και ε, πρόκειται να υπάρξει μία συζήτηση η οποία θα επηρεάσει αποφασιστικά το τελικό πρόγραμμα ε, εναπόθεσης πυρηνικών αποβλήτων στη Γαλλία. Όσον αφορά το σύστημα εναπόθεσης είναι δύσκολο, όπως είπε ο κύριος Άπελ, ε, είναι δύσκολο να υπάρχει διαφάνεια στις διεργασίες αυτές και ιδίως από πλευράς τεχνικής. Γι' αυτό και πιστεύω ότι πρόκειται για κάτι το οποίο πρέπει να ενισχύσουμε ε, εάν ε, υπάρχει ήδη εμπειρία από επιτυχή προγράμματα τα οποία έγιναν αποδεκτά. Ε, το χρονοδιάγραμμα για μια χώρα η οποία δεν έχει μεγάλη πυρνική δραστηριότητα αν κοιτάξουμε τη Φιλανδία μπορούμε να δούμε ότι αυτή τη στιγμή ε, έχει τέσσερις αντιδραστήρες χτίζουν έναν πέμπτο και άρα αξίζει να δημιουργήσουν ένα σημείο εναπόθεσης πράγμα το οποίο δεν συνεπάγεται υποχρεωτικά ότι όλες οι μικρές χώρες πρέπει να δημιουργήσουν σημεία εναπόθεσης. Χώρες σαν την Ελβετία είναι ανοιχτές για περιφερειακή εναπόθεση αλλά ε, συνεχίζουν εντωμεταξύ το ισχύον ε, εθνικό πρόγραμμά τους. Αποδοχή. Πολύ σωστά είπε ο κύριος Άπελ προηγουμένως safety first. Αυτό προέχει παντού, αυτό ακούμε παντού. Αλλά βέβαια το ερώτημα είναι η ασφάλεια επαρκεί. Και το θέμα γίνεται όλο και πιο ασαφές και είναι πολύ δύσκολο να απαντήσουμε. Δηλαδή μπορούμε από τώρα να προεξοφλήσουμε τι θα γίνει σε 100.000 χρόνια. Μπορούμε να έχουμε κάτι το αποδεκτό και ε, και εδώ παρεμβαίνουν και τα κοινωνικά θέματα. Μία σύντομη παρατήρηση στον κύριο ο, Τσουκαλά ε, ε, όσον αφορά τις εναλλακτικέ πηγές ενεργείας. Νομίζω ότι καλό θα ήταν ε, να ε, εξετάσουμε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα παραγωγής ενεργείας και βάσει ε, της συζητήσεως για την αποδοχή και για τα σημεία εναπόθεσης θα πρέπει να εξετάσουμε εξετάσουμε και αυτές τις πτυχές διότι ξέρετε ότι ε, υπάρχει σε πολλές χώρες για οικονομικούς λόγους ε, ε, μια διακοπή των προγραμμάτων πυρηνικής παραγωγής ενεργείας. Ε, θα ήθελα τώρα να παρακαλέσω τον επόμενο μιλητή να παρέμβει ε, όσον αφορά την μεταστοιχείωση και πού βρισκόμαστε, πόσο θα διαρκέσει και τι κοστίζει, ποιος θα το χρηματοδοτήσει. Ε, καταρχήν, πιστεύουμε ότι πρέπει κανείς να διαχωρίσει μεταξύ του partitioning και της μεταστοιχίωσης. Θα αναφερθώ εις ε, ε, το partitioning όπου ε, πιστεύω ότι εδώ αναφερόμαστε εις ε, τα διάφορα στοιχεία και πρέπει ε, να έχουμε υπόψη μας τον κίνδυνο μεταδόσεως. Υπάρχει μία διαδικασία και από το, τη φάση της εργαστηριακής παρακολουθήσεως πρέπει να περάσουμε στην εφαρμογή όπου προχωρούν καλύτερα οι Γάλλοι ε, και ε, το 2012 θα μπορούν να παράγουν αυτό, ε, αυτά τα αποτελέσματα και για ποσότητες ενός κιλού και πιστεύουμε ότι αποτελέσματα αυτά θα έχουμε το 2015 με 2020. Όσον αφορά τώρα τη μεταστοιχείωση. Ε, αφενός πρόκειται για την ε, φυσική διαδικασία η οποία έχει ενισχυθεί αλλά χρειάζεται ακόμη επεξεργασία υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία θα έπρεπε να γνωρίζουμε επακριβέστερα ε, για να μπορέσουμε να τα χρησιμοποιήσουμε σε αντιδραστήρια δηλαδή πως τα ουδετερόνια επί επηρεάζουν τα ακτινίδια και όσον αφορά τη διαδικασία πρέπει να δούμε πόσο από την ε, ισχύουσα τεχνολογία θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε ε, εις ε, τους αντιδραστίες ταχύων νετρονίων δηλαδή πόσο θα μπορέσει με τα καύσιμα τα οποία γνωρίζουμε ε, το πλουτόνιο και ε, να χρησιμοποιήσουμε νέες μορφές ε, με ε, ε, νετρόνια και ακτινίδια. Βεβαίως όλα αυτά ακόμη ε, δεν έχουν προχωρήσει πέραν του εργαστηρίου και δεν χρησιμοποιούνται σε ενεργειακές εγκαταστάσεις οπότε θα πρέπει να αναπτυχθούν για μονάδες 50 έως 100 ΜΒ η Βέλγια η κυβέρνηση είναι η πιο προηγμένη σε αυτόν τον τομέα, δηλαδή ε, είναι έτοιμη να χρηματοδοτήσουν 40% μια τέτοια εγκατάστασης όπου θα προσκαλέσουν και άλλους εταίρους να συμμετάσχουν και εκεί πρέπει να δούμε αν υπάρχει ε, προθυμία εκ μέρου των άλλων κρατών. Αλλά αν λάβω υπόψη μου αυτό το Βέλγιο, ε, βέλγικο πρόγραμμα πρέπει πρέπει να πω ότι είναι μία μονάδα για επίδειξη, όχι για τεχνική εκμετάλλευση και ε, μιλάμε για ένα χρονικό πλαίσιο 10 ετών, οπότε για να μπορέσει να λειτουργήσει επιχειρησιακά θα χρειαζόμαστε να έχουμε ε, πείρα, να παρακολουθήσουμε την ε, βαθμιαία μεταλλαγή του καυσίμου κατά τρόπον, ώστε μετά να μπορέσουμε να επέμβουμε τεχνικά και να δούμε τι γίνεται. Πόσο χρόνο θα διαρκέσει αυτή η διεργασία. Όπως είπα, πολύ αισιόδοξα πιστεύω ότι η βάση απόφασης εάν μία τέτοια εγκατάσταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ε, για μία εθνική αποδόμηση δεν θα επιτευχθεί πριν από το 2030 και Επιπλέον υπάρχει το θέμα της χρηματοδότησης, διότι η διαδικασία αυτή ενεργειακά είναι θετική. Δηλαδή αυτό σημαίνει και αυτό προσπαθούμε να διαπιστώσουμε τώρα, το κόστος μπορεί να επιτευχθεί από την ανάκτηση ενεργείας από αυτή τη διαδικασία κατά τρόπον ώστε να χρηματοδοτήσει την προσπάθεια. Και στη συνέχεια θα πρέπει να εξετάσουμε ορισμένα στοιχεία διότι υπάρχει πολύ ενέργεια και στο πλουτόνιο και εις ε, τα νετρόνια και τα ακτινίδια ε, που θα χρειαστεί να προστατευτεί και είναι και αυτό ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να συνυπολογίσουμε. Πιστεύω όμως και αυτό είναι ο υπολογισμός τον οποίο καταλήγω ότι όσον αφορά τη μεταστοιχείωση πρέπει να γίνουν μεγάλες προσπάθειες διότι ότι όπως ελέγχθη πολύ σωστά αυτά διαρκούν πολύ χρόνο. Ε, είναι δηλαδή μια μακριά διεργασία και δεν έχουμε την αναγκαία στήριξη κατά τρόπον ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα. Ε, ο κόσμος βέβαια έχει και άλλες εναλλακτικές λύσεις. Εκτός από την μεταστοιχίαση μπορούμε να δούμε αν άλλες ιδέες ε, μπορούν να οδηγήσουν σε μία σημαντική μείωση των μακροβίων ε, καυσίμων και εδώ πιστεύω ότι η έρευνα όσον αφορά το φάσμα των νετρονίων χρειάζεται να προχωρήσει διότι χρειαζόμαστε για την σχάση αυτήν την ε, ε, ε, αυτό το φάσμα των νετρονίων για να μπορέσει κανείς να κάψει πιο γρήγορα τα μακρόβια καύσιμα και ε, γι' αυτό έχουν ξεκινήσει εργασίες σε αυτό το τομέα από εμάς αλλά και από άλλους και ε, το τρίτο στοιχείο είναι ε, πολύ πιο μακροπρόθεσμα ότι θα μπορούσε κανείς ε, να πάρει την, ε, ε, την πηγή νετρονίων του αντιδραστήρα και να την μεταστοιχειώσει. Προσπαθούμε μέχρι το 2030 να έχουμε προχωρήσει στην έρευνα όλων αυτών των στοιχείων για να μπορέσουμε να τα αξιολογήσουμε συνολικά. Επανέρχομαι τώρα στην ε, εναπόκτηση ε, διότι έχω ασχοληθεί με το θέμα αυτό και με ενδιαφέρει πολύ. Η κατάσταση στη Γερμανία τουλάχιστον ε, είναι αυτή τώρα ότι η επανάκτηση είναι μία διαδικασία διαδικασία η οποία απαιτεί μεγάλη ασφάλεια και όπως είπε και η κυρία Χάρμς έχει ορισμένα νομικά στοιχεία και ε, έχει προϋποθέσεις. Μπορεί να υπάρξει άδεια ανακτήσεως μόνο εάν είναι ασφαλής. Αυτό για το χρόνο λειτουργίας μιας εγκατάστασης. Για τα 500 χρόνια υπάρχει ένα στόχος ο οποίος δεν χρειάζεται αδειοδότηση αλλά πρέπει να δείξει κανείς ε, πώς έχει καταλήξει σε αυτό τον υπολογισμό ε, εναλλακτικές λύσεις. Πιστεύω ότι στη συζήτηση αυτή πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες ε, δεν θα ξεκινήσουν ε, ε, σήμερα ή αύριο αλλά ήδη παρακολουθούν εδώ και χρόνια. Άρα πρέπει να μετατοπιστούμε κατά 30 χρόνια να μιλήσουμε να θυμηθούμε τις συζητήσεις που είχαμε σχετικά με το τον διαχωρισμό και εδώ θα ήθελα να πω στον συνάδελφο Απέλ ότι δεν θα πετάξουμε ε, μία, ένα πολύτιμο λίθο επειδή τον βρήκαμε κάπου αλλού και άρα στη, σε μία διαδικασία έρευνα στην οποία κάνουμε τώρα ε, για να αξιολογήσουμε το πιο κατάλληλο σημείο εναπόθεσης ε, δεν θα μπορέσουμε τεχνικά ε, να αποφασίσουμε εάν το διαμάντι ή ε, το ρουμπίνι είναι το καλύτερο στοιχείο για την αποθήκευση αυτή και άρα οι τεχνικές γνώσεις θα χρειαστεί να βελτιωθούν. Αυτό ήταν ο πρώτος γύρος μας κυρίες και κύριοι. Έχουμε σεβαστεί περίπου το χρόνο μας Ευχαριστώ και τις χρήσιμες παρατηρήσεις, τις απαντήσεις. Πολλά απαντήθηκαν, ποτέ δεν απαντούνται όλα. Θα χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο χρόνο, γι' αυτό θα ήθελα να ε, ευχαριστήσω τους συμμετέχοντες και να παρακαλέσω τους επόμενους να έρθουν ε, στο βήμα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε.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 Ευχαριστώ. Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε γρήγορα κυρίες και κύριοι θα ήθελα τώρα να καλέσω τους επόμενους ομιλητές για τη στρατηγική ε, των πολύ ραδιενεργών ε, ε, τη στρατηγική της διαχείρισης των πολύ ραδιενεργών αποβλήτων να ζητήσω από τον κύριο Πατράκα να λάβει τον λόγο και να σεβαστεί το χρόνο Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχω δύο είδη διαφάνειών. Πρώτα απ' όλα θα αναφερθώ στην πύρα που έχουμε αποκτήσει στην Φιλανδία για την διάθεση των εξαντλημένων πυρηνικών καυσίμων και μετά για τα όσα έχω μάθει από το Nuclear Energy Forum. Για να επανέλθω λοιπόν στο θέμα που μας αφορά, να σας πω πως έχω μία παρουσίαση στην οποία θα σας κάνω μία επισκόπηση για το πώς εφαρμόζεται η διαχείριση αποβλήτων στη Φιλανδία. Πρέπει να σας πω πως έχουμε δύο ε, ε εταιρείες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούν πυρηνικές εγκαταστάσεις και έχουμε και μία τρίτη η οποία αυτή τη στιγμή κατασκευάζει ε, τέτοιου είδους πυρηνικό εργοστάσιο. Τι λέμε διαχείριση αποβλήτων. Να σας πω πως είναι τα χαμηλής και μέσης ραδιενέργειας απόβλητα και έχουμε δύο χώρους ε, εναπόθεσης ε, που ε, δέχονται αυτά τα απόβλητα. Τώρα για τα εξαντλημένα καύσιμα να σας πω πως αποθηκεύονται σε, μια ενδιάμεση, σε έναν ενδιάμεση χώρο αποθήκευσης και η τελική διάθεση γίνεται από την εταιρεία Ποσίβα, που είναι η δική μου εταιρεία, και η οποία είναι η υπεύθυνη για την τελική διάθεση ε, του πυρηνικού αυτού καυσίμου μετά την αποθηκευσή τους. Εμείς ε, συσταθήκαμε το 1995. Βλέπετε ε, ότι το 60% ανήκει στην Τεολισούνεν Βόημα ΟΗ με αποστολή, με αποστολή την ανάπτυξη, αδειοδότηση και εφαρμογή της ασφαλούς διάθεσης ε, του εξαντλημένου πυρηνικού καυσίμου. Αυτή τη στιγμή έχουμε υποβάλει μία αίτηση για να αδειοδοτηθούμε για το 2012 και η εταιρεία μας αυτή τη στιγμή κάνει χωροθέτηση σε υπόγειες εγκαταστάσεις στο «ον καλό» και θα σας εξηγήσω ποια είναι αυτή η εγκατάσταση αργότερα. Σχεδιάζουμε τις μονάδες που θα χρησιμοποιηθούν για την τελική διάθεση και κάνουμε έρευνα και αξιολόγηση της μακροπρόθεσμης ασφάλειας. Η εταιρεία μας αυτή τη στιγμή αναπτύσσει δεξιότητες και δυνατότητες για την εφαρμογή όλων αυτών της τελικής δηλαδή διάθεσης. Έχουμε στο Ολκυλουότο 150 άτομα περίπου προσωπικό, αλλά αν δούμε τι γίνεται με τις υπεργολαβίες που έχουμε, ουσιαστικά απασχολούμε γύρω στα 300 άτομα. Ε, ετήσιος προϋπολογισμός 60 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ θα σας δείξω μια φωτογραφία ε, της, ε, του χώρου στο Όλ Κιλουότο... το καλοκαίρι του 2009. Βλέπετε λοιπόν την ε, υπέργεια άποψη και θα σας δείξω και τι έχουμε ως υπόγειες εγκαταστάσεις. Έχουμε τρεις μονάδες και η απόσταση μεταξύ των δύο εγκαταστάσεων που έχουμε, γιατί σας είπα έχουμε και άλλη μία, είναι γύρω στα 20 χιλιόμετρα, γύρω στα 2 χιλιόμετρα. Έχουμε κάνει προσπάθειες τα τελευταία 40 χρόνια και έχουμε και κάποιες ε, προοπτικές για το μέλλον μέχρι το 2020. Κάνουμε στην Φιλανδία ήδη από την ε, δεκαετία του 70 κάποιες μελέτες βιωσιμότητας για την γεωλογική αναπόθεση. Αποφάσισε μετά η κυβέρνηση ποια θα είναι και θα είναι, ποιοι θα είναι μας στόχη και το χρονοδιάγραμμα για την διάθεση των αποβλήτων και για τα εξαντλημένα καύσιμα και τα ιδιαίτερα ραδιενεργά απόβλητα, ήδη το 1983 η κυβέρνηση αποφάσισε ότι ο χώρος θα πρέπει να επιλεγεί το 2000 έτσι ώστε η διάθεση να ξεκινήσει από το 2010. Για να προχωρήσουμε λοιπόν ε, σύμφωνα με αυτό το χρονοδιάγραμμα χρειάστηκε να προετοιμάσουμε όλο το σχετικό υλικό. Πριν λοιπόν με την προσπάθεια χωροθέτησης ε, για τις περιπτώσεις αυτών των ε, καυσίμων και για τα χαμηλής και μέσης ραδιενεργίας ε, κατασκευάστηκαν τη δεκαετία του 90, επιλέγει δε ο χώρος του 2000. Θα ήθελα λοιπόν να πάμε στην προηγούμενη διαφάνεια. Η απόφαση λοιπόν η αρχηγή ελήφθη από το Κοινοβούλιο και την κυβέρνηση το 2001 και το δόγμα που ακολουθήσαμε είναι γνωστό. Ορίσαμε λοιπόν τον χώρο και πρέπει να σα πω ότι σε αυτή τη διαδικασία καθυστέρησαμε αρκετά. Ξεκίνησε η κατασκευή των εγκαταστάσεων στο Ονκαλό και έγιναν κάποιες έρευνες στο Ολκιλουότο για να επιβεβαιωθεί η χωροθέτηση και οι μελέτες αυτές τρέχουν ακόμα. Η αίτηση για την άδεια ε, την κατασκευαστική άδεια ε, θα υποβληθεί το 2012 και το 2018 θα καταθέσουμε την αίτηση για την άδεια λειτουργίας. Εδώ θα σας δείξω πώς ε, στήσαμε το πρόγραμμα ερευνών για την επιλογή του χώρου. Από το 83 μέχρι το 85 ξεκινήσαμε με τις προσπάθειες εντοπισμού καταλήλων περιοχών. Βρήκαμε τουλάχιστον 100 τέτοιες περιοχές και περιορίσαμε τον αριθμό αυτό με χαρακτηρισμό και μελέτες χαρακτηρισμού ε, σε τέσσερις περιοχές στη Φιλανδία μεταξύ του 86 και του 92 και η τελική επιλογή έγινε το 1993 στο Εουραγιώκη. Ε, η άλλη εγκατάσταση στο Εουραγιώκη επιλέγει το 2000 χρησιμοποιούμε το δόγμα διάθεσης που είναι το KBS 3, το οποίο θα, επιλέξει, θα παρουσιάσει με περισσότερες λεπτομέρειες ο συνάδελφος αργότερα. Δεν θα σας δώσω τώρα τις λεπτομέρειες. Να σας πω πως έχουμε δύο βασικές εναλλακτικές. Έχουμε KBS 3V ε, που είναι κάθετη ε, ε, εναπόθεση και την KBS 3H που είναι η οριζόντια. Πρέπει να σας πω πως στην δεκαετία του 80 η τεχνολογία δεν ήταν τόσο προηγουμένη και πρέπει να σας πω πως πριν από 10 χρόνια η η έκανε μια συμφωνία, υπέγραψε μια συμφωνία με μια σουηδική εταιρεία έτσι ώστε όλες αυτές τις τεχνικές ε, ε, παραμέτρους να τις αναπτύξουμε μαζί. Θα ήθελα να εξηγήσω καταρχήν τι ακριβώς έχουμε στον χώρο ε, στην περιοχή Όγκαλο. Είναι μια εγκατάσταση υπόγεια σε βραχώδη περιοχή και βέβαια επαληθεύσαμε την καταλληλότητα αυτού του χώρου μέσω των ερευνών που κάναμε σε διάφορα βάθη. Είμαστε τώρα στα 400 μέτρα βάθος και τα κάναμε σταδιακά και η τελική επαλήθευση θα γίνει βέβαια στο πραγματικό βάθος εναπόθεσης. Ποιο είναι ο στόχος μας σε επίπεδο σχεδιασμό. Να χρησιμοποιηθεί ε, κατά την κατασκευή και τη λειτουργία της, ε, ε, των εγκαταστάσεων υπόγειας εναπόθεσης. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν θα εξοικονομήσουμε χρόνο και θα είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε την εναπόθεση νωρίτερα από ό,τι περιμέναμε. Υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις για θα πρέπει να σχεδιάσουμε και να κατασκευάσουμε τη μονάδα αυτή σύμφωνα με τις απαιτήσει που έχουν οριστεί για τις πυρηνικέ εγκαταστάσεις. Δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα επίσημα την τελική διάθεση, αλλά αυτή τη στιγμή γίνονται εργασίες ε, στην μονάδα αυτή ε, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις ε, περί λειτουργίας πυρηνικών εγκαταστάσεων και μας ελέγχει η Φιλανδική Ρυθμιστική Αρχή για την Πυρηνική Ενέργεια. Αυτό στο οποίο καταλήξαμε, κάτι το οποίο είχαμε φανταστεί από την αρχή, αλλά βρέθηκε και από τις ερευνές μας, είναι πως αυτή η περιοχή, το όγκαλο, μας δίνει την ευκαιρία να αποκτήσουμε και κάποιες γνώσεις, γιατί όταν μπαίνει κανείς στην πραγματική σειρά εργασιών, τότε μόνο γνωρίζει ποιες είναι οι προκλήσεις που θα ε, χρειαστεί να αντιμετωπίσει υπό πραγματικές συνθήκες. Θα σας δείξω πού βρισκόμαστε τον Νοέμβριο του 2000. Βλέπετε λοιπόν πως υπάρχουν αυτές οι, οι σύραγγες οι οποίες ε, φεύγουν από το, ε, το έδαφος και, μέχρι, και πάνε σε βάθος μέχρι 400 μέτρα. Βλέπετε πως είμαστε στα 426 και δίπλα στη σύραγγα αυτή έχουμε και μια κάθετη, ε, έχουμε κάθετες ε, κάθε τα φρεάτια εξαιρισμού και βλέπετε πως το γκρίζο τμήμα είναι αυτό το οποίο ακόμα δεν έχουμε σκάψει. Όταν τελειώσουμε λοιπόν την εξόριξη και εκεί θα έχουμε φτάσει στο τελικό βάθος. Οπότε βλέπετε πως και στα διάφορα σημεία, στα βάθη που είχαμε φτάσει, μπορέσαμε να κάνουμε διάφορες μελέτες. Εδώ έχουμε μια φωτογραφία από την είσοδο ε, στην εγκατάσταση και εδώ είναι ε, μια εικόνα από τη, μία από τις σύραγγες τις οποίες έχουμε εξορίξει. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, γιατί επαναλαμβάνω θέλουμε να πετύχουμε καταρχήν το τελικό βάθος εναπόθεσης και αφού φτάσουμε τότε μόνο ε, θα τελειώσουμε τα δάπεδα ε, και τα τυχώματα. Εδώ έχουμε και μία εικόνα από ένα από τα φρεάτια που θα χρησιμοποιηθούν. Θέλω να σας δείξω και τις εγκαταστάσεις ε, διάθεσης που θα είναι παρόμοιες με αυτές που βλέπετε εδώ στην εικόνα. Το όγκαλο είναι με μπλε χρώμα και γύρω-γύρω θα δείτε ότι έχουμε μία σειρά σύραγγες γύρω-γύρω από αυτήν την μονάδα, όπου το τελικό βέβαια μήκος όλων αυτών θα εξαρτηθεί και από το νόγκο καυσίμου ε, που θα φτάνει σε εμάς, γιατί έχουμε σκοπό να κάνουμε αναπόθεση ε, καυσίμου από τέσσερις εγκαταστάσεις που θα φτάνουν σε εμάς. Δηλαδή, η μονάδα αυτή έχει τη δυνατότητα να διευρυνθεί, αλλά υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί γιατί είναι νησί και δεν θέλουμε ε, να σκάψουμε κάτω από τη θάλασσα. Υπάρχει λοιπόν ένας γεωγραφικός περιορισμός που πρέπει να λάβουμε υπόψη βλέπετε πως αυτές οι σύραγγες δεν είναι ομοιόμορφες και έχουμε και κάποια σημεία κάτω από τα οποία δεν έχουμε σκάψει ε, λόγω ε, της ε, σύστασης των βράχων ορισμένοι δεν έχουν την απαραίτητη σκληρότητα ώστε να σκάψουμε εκεί. Έχουμε κάνει 50 50 γεωτρήσεις ε, για να ελέγξουμε την ποιότητα των πετρωμάτων και έχουμε και ένα τριδιάστατο μοντέλο που δοκιμάζουμε για να εξετάσουμε την αντοχή τους. Για να δούμε λοιπόν τον ε, τελικό προϋπολογισμό, τον οποίο ε, υπολογίζουμε κάθε τόσο. Εδώ έχουμε τον ε, τελευταίο από το 2009. Βλέπετε πως 3 δις ευρώ είναι ο τελικός προϋπολογισμός. Έχουμε τις επενδύσεις που θα γίνουν υπέργεια, που είναι γύρω στα 160 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή είναι οι εγκαταστάσεις που θα τοποθετήσουμε εκεί για τη συσκευασία και τα περιβλήματα. Έχουμε τις επενδύσεις για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε υπογείως. Έχουμε το κόστος λειτουργίας υπέργειο και υπόγειο που λαμβάνονται υπόψη για τα δοχεία και τις δεξαμενές όπως επίσης και το κόστος αποξύλωσης ε, και παροπλισμού. Φτάνουμε λοιπόν σε ένα κόστος 2 δις ευρώ Καταλαβαίνετε λοιπόν πως για τον πετονίτη το κόστος για την κατασκευή των περιβλημάτων δοχείων και δεξαμενών είναι αρκετά υψηλό. Πάντως οι εγκαταστάσεις αυτές θα λειτουργούν για τουλάχιστον 100 χρόνια με αποτέλεσμα τουλάχιστον να προχωρήσουμε ε, σε μια απόσβεση του κόστους επένδυσης. Να πω μόνο πως στη Φιλανδία Έχουμε ένα ταμείο ε, κρατικό διαχείρισης αποβλήτων πυρηνικών. Καταλαβαίνετε λοιπόν όμως πως το κόστος είναι για την τελική διάθεση ε, αυτών των ε, ακτινοβολημένων ή εξαντλημένων καυσίμων είναι τεράστιο. Έχουμε τις δύο εταιρείε που όπως σας επαναλαμβάνω, που όπως σας ανέφερα προηγουμένως έχουν ε, καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες ρεδιενεργών αποβλήτων. Μπορούμε τώρα όμως να περάσουμε στην επόμενη διαφάνεια. Είναι δύσκολο να το δείτε στην οθόνη, είναι πολύ μικρό το μεγεθός της. Εδώ όμως θα σας δώσουμε μια ιδέα για τα διάφορα βήματα στα οποία προχωρούμε. Πρώτα απ' όλα λοιπόν έχουμε τους πυρηνικούς αντιδραστήρες οι οποίοι λειτουργούν και τον κύκλο ζωή τους. Αυτή τη στιγμή στο Λόβισα 1 και 2 ε, θα λειτουργούν μέχρι το 2030 περίπου, στο Ολκυλουότο 1 και 2 μέχρι το 2040 και στο Ολκυλουότο 3 που ακόμα δεν έχει ξεκινήσει να λειτουργεί. Εκεί το σχέδιο είναι ένας κύκλος ζωής 60 ε, ετών. Από το 2013 λοιπόν, αν προλάβουμε το χρονοδιάγραμμα, μέχρι το 2073 περίπου. Μετά θα αποξηλωθεί και η διαχείριση των ε, αποβλήτων χαμηλής και μέσης ραδιονέργειας είναι συνεχής, γιατί σας είπα έχουμε χώρους αναπόθεσης ε, αυτή τη στιγμή και απλώς θα διευρυνθούν για να καλύψουν και τις μελλοντικές μας ανάγκες. Στο επόμενο έχω να σας δείξω την ε, αποθήκευση όπου χρειάζεται ε, να κάνουμε μια ενδιάμεση αποθήκευση καθ' όλη τη διάρκεια ε, μέχρι την τελική εναπόθεση και εδώ βλέπετε πότε θα ξεκινήσουν οι, οι λειτουργίες τελικής διάθεσης. Αν ξεκινήσουμε το 2020 όπως προβλέπουμε, η διάθεση του λοβισα 1 1-2 και ολκυλό το 1-2, 1 και 2, αυτή η ενδιάμεση λοιπόν αποθήκευση θα κρατήσει γύρω στα 70 χρόνια, μέχρι το 2070. Άρα λοιπόν η διάθεση του Ολκυλώτο 3 θα ξεκινήσει μόνο αφού έχει κλείσει το θέμα της διάθεσης για τα απόλυτα της προηγούμενες μονάδες. Άρα λοιπόν μιλάμε για 2100, φτάνουμε στο 2120, με συγχωρείτε. Έχουμε εδώ τις μελάτες για τις διαφορετικές αναλλακτικές ε, λύσεις που έχουμε για την διαχείριση που ξεκίνησαν των ε, εξελιγμένων αυτών απολύτων καυσίμων που ξεκίνησαν όταν ε, ξεκίνησε να λειτουργεί το Λοβίσα 1 και 2 και το Ολκυλουότο 1 και 2 στη δεκαετία του 70 η κυβέρνησή μας δεσμεύτηκε σε ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα γιατί είχαμε καταρχήν ε, φόρτωση και μεταφορά καυσίμων στο εξωτερικό που είχε θεωρηθεί ως η καλύτερη λύση. Αυτό έγινε για τα απόβλητα από τη μονάδα Λοβιίσα. Δηλαδή τα στέλναμε στη Ρωσία ε, για μια περίοδο τουλάχιστον 10 ετών. Για την περίπτωση του Ολκυλουότο το πρόγραμμα ε, δεν μπορούσε πλέον να ακολουθηθεί με τον ίδιο τρόπο. Δεν γινόταν να τα στέλνουμε στη Ρωσία και ξεκινήσαμε ε, την σκέψη για τη διάθεση στη Φιλανδία το 2020. Η γεωλογική εναπόθεση στην ε, Φιλανδία έγινε πλέον ε, νόμος το 1994 για όλο το πυρηνικό, όλα τα πυρηνικά απόβλητα και πλέον δεν στέλναμε τίποτα στη Ρωσία. Η απόφαση αρχής το 2001 ανέφερε πως η διάθεση στο όλκυλότο ε, ευθυγραμμίζεται με το γενικότερο κοινωνικό καλό. Άρα λοιπόν παραμένει στη Φιλανδία. Η εταιρεία Ποσίβα έχει φτάσει στο βάθος ε, διάθεσης στο καλό και το μακροπρόθεσμο πρόγραμμά μας που ε, ξεκίνησε ε, με απόφαση το 1983 εξακολουθεί να είναι ενισχύ, θα ξεκινήσει το 2020. Και αν αυτό συμβεί θα ξεκινήσουμε και θα είμαστε οι πρώτοι στον κόσμο που θα κάνουμε τέτοιου είδους διάθεση. Έχω βέβαια και μερικές διαφάνειες ακόμα, τις οποίες δύο-τρεις ε, διαφάνειες ακόμα που θα ήθελα να σας δείξω. Να σας δείξω λοιπόν να αναφερθώ και κάτι που μου ζητήσανε να αναφέρω, ε, γιατί θα ήθελα να σας εξηγήσω τι κάναμε στο φόρουμ για την Ευρωπαϊκή Πυρηνική Ενέργεια. Έχουμε μία υποομάδα για τη διαχείριση αποβλήτων στα πλαίσια αυτού του φόρουμ και η υποομάδα έχει ως σκοπό να προωθήσει στα κράτη-μέλη την διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων και ε, αναλωμένων καυσίμων. Θέλουμε να δώσουμε λοιπόν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές για την επιτυχή ε, διάθεση αυτών των αποβλήτων και να κατανοήσουμε βέβαια πως η διαχείριση αποβλήτων είναι ενδιαφέρει από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Και πρέπει βέβαια να λάβουμε πώς υπάρχουν και διαφορετικοί τρόποι για επιτυχή διαχείριση. Έτσι Λοιπόν, θέλουμε να δούμε και πώς μπορούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσουμε σε μια επιτυχή διάθεση με ε, γεωλογική απόθεση, κάτι το οποίο ε, ξεκίνησε να εξετάζεται με απόφασή μας και κατευθυντήριες γραμμές από την ε, περσινή χρονιά. Εδώ έχουν τα συμπεράσματα και τις συστάσεις. Οι πολιτικές αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν έτσι ώστε να εξασφαλιστεί πως η γεωλογική διάθεση θα εφαρμοστεί χωρίς χρήστε καθυστερήσεις λαμβάνοντας υπόψη ε, την μεγάλη διάρκεια ε, της ε, διάθεσης και της διαχείρισης της διάθεσης, θα πρέπει τα σχέδια για νέους αντιδραστήρες να μην υποβάλλονται χωρίς μια συνολική και αξιόπιστη μελέτη για την διαχείριση των αρδιενεργών αποβλήτων και καυσίμων. Οι πολιτικές ε, αποφάσεις θα πρέπει να μετατραπούν σε ξεκάθαρες διατάξεις στις εθνικές πολιτικές διαχείρισης αποβλήτων και θα πρέπει αυτά να, ε, καθιερωθούν μέσω ενός πλαισίου νομικού το οποίο θα παρουσιαστεί εν ευθέτω χρόνο. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη που σας έκοψα, αλλά θα ήθελα να κρατήσουμε και λίγο χρόνο για τις ερωτήσεις. Ο κύριος Βάν είναι ο επόμενος ομιλητής. 15 λεφτά μου δίνετε. Χα. Λέγομαι Γιώχαντ Σβάν και δουλεύω ε, στην ε, μη κυβερνητική οργάνωση της Σουηδίας για, την, ε, για τα πυρηνικά απόβλητα. Ε, θέλω να σας πω κάποια πράγματα για το πώς διαχειριζόμαστε τα πυρηνικά απόβλητα στην Σουηδία. Ευχαριστώ την Επιτροπή σας που μου έδωσε το, την ευκαιρία να μιλήσω για αυτό το θέμα. το γραφείο, το σουηδικό της μη κυβερνητικής αυτής οργάνωσης, είναι μια οργάνωση που υποστηρίζεται από τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική με κυβερνητική οργάνωση της Σουηδίας για τη διατήρηση της φύσης και ασχολείται με θέματα πυρηνικών αποβλήτων. Ε, λαμβάνουμε χρηματοδότηση για να συμμετέχουμε στη διαδικασία ε, διαβούλευσης για τη δημιουργία ενός χώρου εναπόθευσης για τα αναλωμένα πυρηνικά κάψιμα ε, του πυρηνικού εργοστασίου Forsmark. Ε, Υπάρχει μια ειδική εταιρεία, η SKB, υπεύθυνη για την διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων, που την, ε, το Μάρτιο του 2011 θα υποβάλει μια αίτηση ε, για να πάρει άδεια ένας χώρος εναπόθεσης. Ε, μιλάμε για ένα project 30 ετών. Ε, βρισκόμαστε στην ακτή της Βαλτικής, περίπου 100 χιλιόμετρα βόρεια από τη Στοκχόλμη, κοντά ε, στο εργοστάσιο Forsmark. Ε, έχει γίνει μια διαδικασία διαβούλευσης πριν από την υποβολή της αίτησης και έχουμε, έχουν συζητηθεί διάφορα θέματα. Ε, καταρχάς πόσο εξασφαλίζουμε την ασφάλεια μακροπρόθεσμα. η διαδικασία αδειοδότηση θα κρατήσει κάποια χρόνια και εκεί θα εξεταστούν διάφορα θέματα. Φυσικά είναι μεγάλη πρόκληση να βρούμε έναν τρόπο διαχείρισης των μακρόβιων και επικίνδυνων πυρηνικών αποβλήτων από τα, τις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Καταρχάς ε, η ραδιενέργεια. Θα πρέπει να απομονώσουμε αυτά τα απόβλητα από τον άνθρωπο και το περιβάλλον για εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια. Ε, μην ξεχνάμε ότι το πλουτόνιο που, μπορεί, που παραμένει στα αναλωμένα πυρηνικά καύσιμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πυρηνικά όπλα. Ε, επίσης, ε, το πιο σημαντικό ισότοπο του πλουτονίου έχει χρόνο ζωή 24.000 χρόνια. Ε, και επομένω θα πρέπει ε, να εποπτεύουμε αυτά τα πυρηνικά απόβλητα για πάνω από 100.000 χρόνια. Επίση, υπάρχει και χημικό κίνδυνο. Ε, μπορεί να έχουμε δηλαδή βαρέα μέταλλα ε, και, άλλα, και άλλες ουσίες που είναι επικίνδυνες. Με βάση τον νόμο της Σουηδίας, η πυρηνική βιομηχανία είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων μας. Θα πρέπει να βρούμε μία βιώσιμη μέθοδο για την τελική εναπόθεση των αποβλήτων με αυστηρά κριτήρια για τη μακροπρόθεσμη ασφάλεια, όπως λένε και οι ρυθμιστικές αρχές. Έχει δημιουργηθεί ένα οικονομικό σύστημα για να εξασφαλίσουμε ότι ισχύει η αρχή του ορυπαίνων πληρώνει. Για κάθε κιλοβατόρα που παράγουμε ε, ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή, θα πρέπει η πυρηνική βιομηχανία να πληρώνει ένα τέλος. Ε, υπάρχει λοιπόν ακριβώ μια ειδική εταιρεία η οποία έχει το, το καθήκον ακριβώς να διαχειριστεί τα πυρηνικά απόβλητα. Τη λέμε SKB. Στη Σουηδία τα αναλωμένα πυρηνικά καύσιμα διατίθενται σε ένα γεωλογικό χώρο εναπόθεσης ε, χωρίς ε, επανεπεξεργασία. Ήδη ξεκινήσαμε τη διαδικασία, τη διαδικασία από την δεκαετία του 80. Η εταιρεία αυτή SKB εδώ και 30 χρόνια προσπαθεί να βρει ένα κατάλληλο χώρο απόθεσης. Έχει δημιουργήσει τη μέθοδο KBS. Έχουμε φτάσει στην, στο στάδιο SBS 3. Είναι η ίδια μέθοδος που χρησιμοποιούν και στη Φιλανδία για το δικό τους χώρο εναπόθεσης. Και είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι η Φιλανδία βασίζεται αποκλειστικά στην ανάλυση για την ασφάλεια που θα κάνουμε εμείς στη Σουηδία. Και πιστεύω ότι δεν μπορούν να προβούν στο, στο δική τους εναπόθεση αν εμείς δεν του δώσουμε το τελικό πράσινο φως μετά την διαδικασία της αντιοδότησης. Θα εξετάσουμε αυτή τη μέθοδο KBS Υπάρχουν διάφορα περιβαλλοντικά θέματα που θα εξεταστούν στη διαδικασία διοδότηση, αλλά καταρχά να σα εξηγήσω ποιο είναι το σουδικό ε, σύστημα για τη διαχείριση των αποβλήτων. Ε, για τα χαμηλά, α, χαμηλές απόβλητα, ε, τα απόβλητα από ξενοδοχή, από νοσοκομεία και τη βιομηχανία κτλ. Ε, έχουμε μια εγκατάσταση, την SFR, ε, που έχει οικοδομηθεί κοντά ε, στο πυρηνικό εργοστάσιο, κάνουμε τη ε, μεταφορά των αποβλήτων με πλοίο. Ε, αυτό το χώρο αναπόθεση SFR βρίσκεται 60 μέτρα κάτω από τη θάλασσα. Και μιλάμε για μια λειτουργία πάνω από 500 χρόνια. Ε, υπάρχουν κάποιες σύραγγες, βάζουμε αυτά τα απόβλητα σε, σε αποθήκες, σε σάιλο. Βλέπετε την εικόνα ε, χρησιμοποιούμε αυτά τα τούνελ σε περίπτωση που κλείνουμε κάποιου ειδικού αντιραστήρε. Τα αναλωμένα ε, καύσιμα από τα ε, εργοστάσια μας πηγαίνουν σε μια κεντρική εγκατάσταση, προσωρινή εγκατάσταση, το κλαμπ. Αυτό το κλαμπ βρίσκεται 75 μέτρα κάτω μέσα στο βραχώδη πέτρωμα, βραχώδες πέτρωμα και όλα τα αναλωμένα ε, καύσιμα από τις σουηδικές εγκαταστάσεις βρίσκονται εκεί. Επομένως καταλαβαίνετε ότι εδώ υπογείως υπάρχει μεγάλη δραστηριότητα. Στα επόμενα βήματα ε, η εταιρεία SKB θα κατασκευάσει, θα κάνει μάλλον μία αίτηση για να κατασκευάσει ένα τελικό χώρο αναπόθεσης για τα αναλωμένα καύσιμα η άδεια θα αφορά και μια εγκατάσταση για τη δημιουργία περιβλημάτων, όπου μπορούμε να βάζουμε σε δοχεία τα, τα απόβλητα αυτά. Θα επανέλθω στα δοχεία αυτά, γιατί είναι πολύ σημαντικό θέμα για την ασφάλεια της μεθόδου αυτής ε, KBS. Αυτή η μέθοδος για τα απόβλητα υψηλής αδιενέργειας ξεκίνησε από τη δεκαετία του 70. Ε, και στα μέσα της δεκαετίας του 70 έγιναν πολλές προσπάθειες. Πάνω από 30 χρόνια λοιπόν ε, έχει πίσω της αυτή η μέθοδο. Το 83, όπως βλέπετε στο, στη διαφάνεια, ε, ξεκινήσαμε με αυτή την εγκατάσταση. Η βασική ιδέα στη μέθοδο KBS είναι να κατασκευάσουμε ένα γεωλογικό χώρο εναπόφεσης 500 μέτρα μέσα στο πετρόδες ε, στο βράχο, ε, κατασκευάζουμε σύραγγες. Τώρα, πώς εξασφαλίζουμε την ασφάλεια. Έχουμε κάποια ε, τεχνητά φράγματα από δοχή, από χαλκό, που περιβάλλονται από ένα α, δηλαδή που είναι ένα είδος αργύλου. Ε, υπάρχει πρόβλημα με τη διάβρωση όμως, δηλαδή μπορεί να σκουριάσουν αυτά τα ε, ε, δοχεία και αυτό μπορεί να συμβεί μέσα σε 100.000 χρόνια. Το βασικό θέμα είναι ε, να μην φτάσει το νερό σε αυτά τα δοχεία χαλκού. Όποιος παρατηρεί βλέπει... Θα θυμάται και την προηγούμενη παρουσίαση που έκανε ο κύριος Πετράκα για το δικό τους χώρο εναπόθεσης, ε, που αντέγραψαν το δικό μας μοντέλο το φιλανδικό μοντέλο εξαρτάται αποκλειστικά από το κατά πόσον θα εγκριθεί το δικό μας, η δική μας αίτηση δηλαδή στη Σουηδία. Πριν κλείσω ε, και μπω θα μπω στα περιβαλλοντικά θέματα, αλλά πρώτα θα μιλήσω για την επιλογή του χώρου. Είχαμε πάρα πολλές αποτυχίες, αλλά μετά από πολλά χρόνια η εταιρεία SKB έκανε κάποιες έρευνες σε δύο τόπους που βρίσκονται παρακείμενοι στο πυρηνικό εργοστάσιο. Ένα στο Σκασάμ και ένα στο ΦΟΡΣΜΑΡΚΑ. Τον Ιούνιο του 2009 ε, επελέγει ε, από την εταιρεία το ΦΟΡΣΜΑΡΚΑ. Ε, επίσης θα χτιστεί και ένα εργοστάσιο στο Σκασάμ ε, που θα ασχολείται με την κατασκευή των περιβλημάτων των ε, αποβλήτων. Η SKB είπε δημόσια ότι σκοπεύει να υποβάλει μια ε, αίτηση για να λάβει άδεια για την ε, μέθοδο KBS για ένα χώρο ε, εναπόθεσης το Μάρτιο 16 Μαρτίου του 2011. Θα υποβληθεί στις ρυθμιστικέ αρχές τη Σουηδική Αρχή Πυρηνική Ασφάλειας με βάση το νόμο για τα πυρηνικά και στο, και στο περιβαλλοντικό δικαστήριο με βάση το περιβαλλοντικό νόμο. Λοιπόν, η αίτηση αυτή θα δώσει στις ρυθμιστικές αρχές να ζητήσω μία σειρά από στοιχεία, παραδείγματο χάρη αποτελέσματα από έρευνε που έχουν κάνει για το κατά πόσο δεν υπάρχει πρόβλημα με τη διάβρωση. Ε, θα ολοκληρωθεί η διεκπαιρέωση της ε, αίτηση μέσα σε τρεις μήνες. Και οι ρυθμιστικές αρχές θα μας πούν την άποψή τους για, το, για τη μέθοδο αυτή και ABS. Η όλη διαδικασία για την αδειοδότηση θα μας πάρει περίπου τρία χρόνια. Και το και οι ρυθμιστικές αρχές και το δικαστήριο θα δώσει συστάσεις στην κυβέρνηση, αλλά η κυβέρνηση θα αποφασίσει αν θα δώσει την άδεια ή όχι. Η απόφαση ε, αποκλείεται να, να ληφθεί πριν από το 2014, το νωρίτερο το 2014. Υπάρχουν τώρα πολλά περιβαλλοντικά θέματα και ανησυχίες τα οποία θα πρέπει να εξεταστούν στη διαδικασία αδειοδότησης. Ε, ένα τελικός χώρος διάθεσης για αυτά τα αναλωμένα καύσιμα δεν πρέπει να, από αυτόν δεν πρέπει να εκλείεται ραδιενέργεια για μια περίοδο 100.000 χρόνια. Ε, μια τέτοια αναπόθεση στα 500 μέτρα στη Σουηδία ε, μπορεί να δημιουργεί προβλήματα διάβρωσης από τα υπόγεια νερά το βασικό θέμα είναι λοιπόν να έχουμε φραγμούς από άργυλο και από χαλκό για να απομονώσουμε ακριβώς αυτό το χώρο από το περιβάλλον. Ε, δεν ξέρουμε όμως πώς θα συμπεριφερθεί ε, το χημικό και βιολογικό περιβάλλον μακροπρόθεσμα ε, και πώς θα αντέξουν αυτά τα τεχνικά φράγματα χαλκού και αργύλου. Ε, δεν μπορούμε να το προβλέψουμε αυτό και διάφορα θέματα ε, δεν μπορούμε να τα αποφασίσουμε. Η μέθοδος KBS βασίζεται σε ένα μοντέλο δεν ξέρουμε τώρα το το μοντέλο αυτό αν είναι πλήρες ή όχι, είναι συζητήσιμο. Το πιο σημαντικό είναι ότι γίνεται μια συζήτηση στη Σουηδία και διεθνώ τα τελευταία χρόνια ε, για την υπόθεση ότι ο χαλκός στα δοχεία είναι υποτίθεται αδρανής στη διάβρωση ε, γύρω σε σχέση με το περιβάλλον. Αλλά δεν έχει επιλύθει αυτό το θέμα. Αυτό είναι ερωτηματικό ανοιχτό. Ε, το θέμα της διάβρωσης του χαλκού είναι ένα θέμα προς Στη Σουηδία αναμένεται ότι τα επόμενα 100.000 χρόνια θα υπάρξουν διάφορες περιοχές, ε, εποχές παγετώνων. Και οι παγετώνες αυτοί θα οδηγήσουν σε μεγάλες διακοιμάσεις στο χημικό και βιολογικό περιβάλλον που θα επηρεάσει αυτά τα φράγματα που δημιουργούν, που φτιάχνουν οι άνθρωποι. Το ίδιο θέμα τίθεται και στη Φιλανδία βεβαίως και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Ε, στα μοντέλα που φτάνουμε για το χώρο διάθεσης, για το χώρο εναπόθεσης, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, ε, λάβουμε, λαμβάνουμε υπόψη μας μάλλον, ότι μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα των 100.000 χρόνων θα έχουμε μάλλον τρεις εποχές ε, παγετώνων. Οι παγετώνες αυτοί θα επηρεάσουν και φυσικά το χώρο εναπόθεσης, ε, πλευρικές ε, μετακινήσεις, ε, σεισμοί, μόνιμη μόνιμο πάγο στα πετρώματα κτλ. Επομένω, υπάρχουν πολλέ αβεβαιότητε για την μακροπρόθεσμη φυσική, χημική και βιοχημική συμπεριφορά ε, του χώρου εναπόθεσης και η διαδικασία διοδότησης θα δείξει αν οι ρυθμιστικές αρχές ε, και οι υπόλοιποι συμφωνούν ε, και θεωρούν ότι υπάρχει υπαρκής ασφάλεια. Και να μην ξεχνάμε ότι τα αναλωμένα καύσιμα περιλαμβάνουν, περιέχουν πλουτόνιο, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να παραχθούν πυρηνικά όπλα Κίνδυνο που δημιουργείται για τα επόμενα 100.000 χρόνια. Επομένω ε, είναι ένα θέμα που πρέπει να το παρακολουθούμε ει το δίνεκε. Τώρα πάμε στη διαδικασία της αδειοδότηση. Καταρχάς, θα υπάρξουν κάποια νομικά θέματα βεβαίως. Η αρχή ε, για την ασφάλεια από τη ραδιενέργεια θα πρέπει να ασχοληθεί με το αν η διαδικασία διαβούλευση ήταν σωστή, αν διενεργήθηκε με το σωστό τρόπο και αν τηρούνται τα οι νομικές προδιαγραφές. Ε, επίσης, ε, αυτό το μοντέλο ε, αντέχει στον έλεγχο σε μακροπρόθεσμη ανάλυση. Αυτά τα σενάρια για τις εποχές των παγετών καλύπτονται με το σωστό τρόπο. τι θα γίνει με τα σενάρια για έκκληση ραδιενέργειας. η SKB μπορεί να αποδείξει ότι το σημαντικό θέμα του αργύλου δεν θα υποστεί διάβρωση κατά τη διάρκεια των παγετώνων. Επίσης, όλα τα στοιχεία που βάζουμε στο μοντέλο θα πρέπει να επαληθεύονται. Το θέμα είναι, καταρχάς, τι γίνεται με τα πρώτα χίλια χρόνια στο χώρο εναπόθεσης. Να μην ξεχνάμε ότι δεν υπάρχουν επαρκή πειραματικά στοιχεία που υποστηρίζουν την ιδέα ότι ο χαλκός δεν διαβρώνεται στο περιβάλλον αυτό του χώρου εναπόθεσης. Θεωρητικά υπάρχει μια θεωρία που υποστηρίζει ότι δεν διαβρώνεται, αλλά πειραματικά δεν το έχουμε αποδείξει αυτό. Το πρόβλημα της διάβρωσης θα γίνει χειρότερο στην αρχή όταν ο χώρος αναπόθεσης τα πρώτα χιλιά χρόνια είναι θερμός. Επίσης, το θέμα είναι αν ο άργυλος θα φουσκώσει και θα συμπεριφερθεί όπως προβλέπεται, κάτι που το επιθυμούμε. Η SKB έχει πολλά προβλήματα με τα αποτελέσματα της έρευνας στο χώρο του, της συναπόθεσης. Ορισμένοι ανεξάρτητοι ερευνητέ θεωρούν ότι θα υπάρξουν πολλά προβλήματα διάβρωση τα πρώτα χίλια χρόνια. Άλλα θέματα για την αδειοδότηση αφορούν την διείσδυση, ε, τον κίνδυνο ανάκτηση και επομένω ε, μακροπρόθεσμη παρακολούθηση ει ε, κίνδυνος ε, με πρόθεση χωρίς πρόθεση. Ε, και αυτό θα πρέπει να το δούμε σε συνδυασμό με την ανάκτηση. Ε, επίσης θα πρέπει να παρακολουθούμε το πλουτόνιο γιατί υπάρχουν κίνδυνοι για τη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Επίσης, με βάση τον περιβαλλοντικό νόμο της ε, Σουηδίας θα πρέπει να υπάρξουν παρουσιαστεί όταν κάνει κανείς κάποια αίτηση και εναλλακτικού χώρου εναπόθεση. Θα πρέπει να δείξουμε δηλαδή ότι ο χώρο που επιλέξαμε ε, επιλέγει με το σωστό τρόπο και ότι είναι ο κατάλληλο χώρο. Βέβαια, το δικαστήριο θα αποφασίσει ποιο είναι ο καλύτερο χώρο, αλλά υπάρχουν διάφορα θέματα που υπησέρχονται εδώ. Η SKB επίση πρέπει να δείξει ότι έχει, κάνει, ε, έχει μελετήσει εναλλακτικέ μεθόδου με τον καλύτερο τρόπο. Υπάρχουν άλλε εναλλακτικέ. Ε, Παραδείγματος χάρη έχουμε συζητήσει μία άλλη μέθοδο ε, των βαθιών γεωτρήσεων που μπορεί να είναι πιο ασφαλός, ασφαλής ε, περιβαλλοντικά και μπορεί να μην δημιουργεί προβλήματα με την ε, δίσδυση. Είτε με πρόθεση είτε από πρόθεση. Επομένως τελικά, πού είναι τα μείζωνα προβλήματα. τι γίνεται, τι θα γίνει αν ε, δημιουργεί πρόβλημα με τη διαδικασία διοδότησης και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στη Σουηδία όπως είχαμε προβλέψει. Παρότι οι εξελίξεις δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια, μπορεί να υπάρξουν σοβαρά προβλήματα για την εταιρεία ε, KBS. Ε, δεν είναι δεδομένο ότι η εταιρεία αυτή θα πάρει την άδεια αν τα θέματα της διάβρωσης του χαλκού ε, των δοχείων ε, δεν έχουν λυθεί, τότε είναι δυνατόν η εταιρεία SKB να τροποποιήσει τη μεθοδό της. Ε, η ιδέα των ε, εμποδίων, των φραγμών που κατασκευάζει ο άνθρωπος θα πρέπει να εγκαταληφθεί. Επίσης, με βάση το σύστημα KBS Θα πρέπει να δούμε ε, αν ε, αυτή η φραγμή που τους φτιάχνει ο άνθρωπος, αυτά εμπόδια, ε, είναι ασφαλή μακροπρόθεσμα και μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε σε οποιοδήποτε πέτρωμα. Η μέθοδος KBS θα επηρεάσει σίγουρα και τη Φιλανδία, τον Καναδά, το Ηνωμένο Βασίλειο, τα δικά του συστήματα διαχείρισης, όπου προβλέπουν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη μέθοδο KBS. Όσοι θέλουν περισσότερες πληροφορίες, ε, έχουμε την, ε, το site μας εδώ, www.mkg.se. Ε, οι μυστικές αρχές έχουν αυτή το site www.ssm.se και ο χώρος, το site της εταιρείας είναι www.skb.se. Βεβαίω έχω ετοιμάσει και κάτι αντίτυπα, τα οποία μπορείτε να πάρετε αν σα ενδιαφέρει η δουλειά μα. Αυτά. Τελειώνει εδώ η παρουσίασή μου. Σα ευχαριστώ. So, last but not least... Ε, ε, τελευταίος. ο κύριος ε, Ντένις Χιούγκελμαν, αντιπρόεδρος της Αρέβα. Καλημέρα σας. Okay. <laughs> Sorry. Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν με τις διαφάνειες, ήμουνα λίγο βιάστηκα λοιπόν πολύ. Πριν μπούμε κατευθείαν λοιπόν στο θέμα της ανακύκλωσης, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας το τι ακριβώς διακυβεύεται όταν μιλάμε και τι ακριβώς σημαίνει πυρηνική, πυρηνικά απόλυτα. Στη Γαλλία, να, ένα θαυμάσιο παράδειγμα, γιατί ξέρετε πως η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι κυρίως πυρηνική στη Γαλλία. Στη Γαλλία λοιπόν έχουμε ε, πολύ ραδιοενεργά απόβλητα. Έχουμε 10 γραμμάρια ανά 20 με 30 ε, γραμμάρια ε, μακρόβιου αποβλήτου. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε πως την αιωνιότητα εμείς θα καλύψουμε με ε, τα απόβλητα που παράγουμε, άρα λοιπόν είναι απαραίτητο να τα ανακυκλώνουμε. Τι ακριβώς σημαίνει πυρηνικό καύσιμο. Έχω εδώ λοιπόν ε, μια πολύ ένα πολύ κλασικό παράδειγμα με τι περιεχόμενο όταν αυτό φτάνει στην ε, ε, πυρηνική εγκατάσταση, γύρω λοιπόν στα 5 κιλά ουρανίου για να προχωρήσει σε παραγωγή ηλεκτρική ανέργεια. Τέσσερα χρόνια λοιπόν χρησιμοποιείται και στο τέλος το εξαντλημένο καύσιμο έχει περιεκτικότητα 95% ουρανίου, 1% πλουτονίου, το οποίο ε, κατασκευάστηκε στον πυρηνικό πυρήνα κατά τη διάρκεια της, ε, ε αλυσίδας, ε, ε, πυρηνικής χάσης και μιλάμε δηλαδή για ένα 4% προϊόντων όταν μιλάμε για ανακύκλωση, μιλάμε για ανακύκλωση του 96% των πρώτων υλών. Μιλάω λοιπόν για ανακύκλωση ουρανίου και πλουτονίου. Πώς μπορεί να συμβεί αυτό. Μπορεί να το κάνουμε. Ε, συλλέγουμε τα αναλωμένα καύσιμα από τους πελάτες μας και αυτά τα ανακυκλώνουμε. Κάνουμε μία αναδιαχωρισμό ουρανίου και πλουτονίου και αυτό τα συσκευάζουμε, τα απόβλητα ε, των καυσίμων ε, με ένα ε, προϊόν σχάσης το οποίο είναι οι στάχτες ουσιαστικά της πυρηνικής αντίδρασης μέσα στον πυρήνα που συσκευάζονται και από αυτό παράγουμε καινούρια καύσιμα ξανα, ε, τα ξαναεμπλουτίζουμε. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή, ότι μιλάμε για κάψιμα στα οποία ξαναεισάγουμε ουράνιο μέσω του πλουτονίου που είναι ένα εξαιρετικά ραδιενεργό υλικό. Μιλάμε λοιπόν για ενέργεια. Ένα γραμμάριο πλουτονίου είναι το αντίστοιχο ενός τόνου ε, πετρελαίου για την παραγωγή ενέργειας. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε τι ακριβώς έχουμε στις εγκαταστάσεις μας. Μετά στέλνουμε αυτά τα νέα καύσιμα στους πελάτες μας, τα οποία πηγαίνουν στην ε, ενδιάμεση εναπόθεση ή αποθήκευση ως συσκευασμένα απόβλητα. Δεν μιλάμε για σχέδια, μιλάμε για κάτι το οποίο ήδη γίνεται και το οποίο ξεκίνησε τη δεκαετία του 70 εδώ στο Βέλγιο, όπου οι πρώτοι ράδοι καυσίμων χρησιμοποιήθηκαν από τους Βέλγους και αυτή τη στιγμή έχουμε 36 πυρηνικές εγκαταστάσεις που χρησιμοποίησαν ή χρησιμοποιούν αυτήν την τεχνολογία. Και θα σας διαβάσω τις λεπτομέρειες από τη διαφάνεια. Αλλά θα δείτε που πάμε. Ελβετία, Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο. Και εδώ, αν κοιτάξουμε και για το τι σημαίνει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δείτε πως έχουμε και την Ιαπωνία, όπου ε, χρησιμοποιούν αυτήν την ε, ανακύκλωση ε, στις πυρηνικές εγκαταστάσεις σε ένα πυρηνικό εργοστάσιο έχουμε μάλιστα και τέτοιου είδους καύσιμα που χρησιμοποιούνται για κάποιες δοκιμαστικές ε, μελέτες για τη χρήση αυτών των καυσίμων και σε μελλοντικέ εγκαταστάσεις. Εδώ λοιπόν έχουμε 19 αντιδραστήρες με το ERU καύσιμο που χρησιμοποιούν δηλαδή το εμπλουτισμένο καύσιμο ουρανίου το οποίο παράγεται επαναλαμβάνω από ανακυκλωμένα υλικά θα μπω και πιο βαθιά στο θέμα ε, για την επεξεργασία των ε, καυσιμών που κάνουμε και να σας πω επίσης τι κάνουμε κατά τη στιγμή της ανακύκλωσης. Έχουμε λοιπόν την αποδόμηση του καυσίμου Μιλάμε για τα μεταλλικά υλικά, τα οποία δεν περιέχουν καμία ποσότητα πυρηνικού υλικού, ε, που δεν είναι ε, ρηπογόνα, αλλά έχουν έρθει σε επαφή και με τα προϊόντα σχάσης και με το ουράνιο και με το πλουτόνιο κατά τη διάρκεια της χάση στον πυρήνα. Ε, προσπαθούμε λοιπόν να μειώσουμε τον όγκο και αυτό που κάνουμε είναι μία συμπίεση των μεταλλικών αυτών για να μπορούμε μετά να τα ανακυκλώσουμε πιο εύκολα. Η διαδικασία που ακολουθούμε είναι η, η αλοποίηση και να σα εξηγήσω ακριβώς τι είναι. Όλοι γνωρίζουμε πως ο μόλυβος είναι εξαιρετικά τοξικό χημικό. Πολύ χημικό, τοξικό. Και βέβαια εμείς όλοι πίνουμε από ποτήρια, από κρίσταλο και ο κρίσταλο ξέρετε ότι είναι ένας άλλο. ο οποίος δεν οδηγεί όμω σε τοξική δηλητηρίαση από την περιεκτικότητα, γιατί βέβαια όταν πίνετε από το ε, ποτήρι ε, φεύγει στην ατμόσφαιρα. Όταν λοιπόν, λοιπόν για σχάση, η οποία γίνεται μέσα στη μήτρα, τι σημαίνει αυτό. Αν λοιπόν διασπάσει τέτοιο μπλοκ, χωρίζεται σε δύο μπλοκ προϊόν ή άλλου σχάσεις, το οποίο όμως δεν εκπέμπει κανεί στην ατμόσφαιρα. Άρα λοιπόν, στο τέλος των δύο διαδικασιών χρησιμοποιούμε ανοξίδωτα περιβλήματα για να συσκευάσουμε αυτά τα απόβλητα, και πρέπει να σας πω πως το η εξωτερική μορφή και το σχήμα συμπίπτει απόλυτα με το καύσιμο το οποίο περιέχει. Άρα λοιπόν αυτές οι κάσκες ή δοχεία μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν και αυτό διευκολύνει τις διαδικασίες και στην αποθήκευση αλλά και στην μελλοντική εναπόθεση σε μεγάλο βάθος. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτό το καθολικό δοχείο, το οποίο έχει αδοδιοτηθεί σε διάφορες χώρες και βλέπετε τις χώρες με πορτοκαλί, στις οποίες έχει λάβει την άδεια, είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, κάτω χώρες, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ελβετία, η Γαλλία και η Ιαπωνία που βλέπετε δεξιά εκτός Ευρώπης και στη διαδικασία διαδιοδότησης βρισκόμαστε στην Ιταλία, στην Αυστραλία και στην Ισπανία. Γιατί βέβαια εμείς ανακυκλώσαμε και κάποιο ερευνητικό και καύσιμο από ερευνητικούς αντιδραστήρες από την Αυστραλία. Λοιπόν, αυτό το δοχείο σήμερα είναι το στάνταρ το οποίο χρησιμοποιούμε και το οποίο χρησιμοποιούν και οι συνάδελφοί του Σέλαφιλτ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εδώ πρέπει να προσθέσω πως όλα αυτά τα δοχεία δεν περιέχουν πια ε, σχάσιμο υλικό, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως εμείς θα μειώσουμε το επίπεδο ασφαλείας, γιατί Μπορούμε βέβαια να τα αποθηκεύσουμε και τελικά πρέπει να σας πω ότι δεν περιέχουν καθόλου πλουτόνιο. Όμως, σε σχέση με την άμεση εναπόθεση, δηλαδή στην άμεση απόθεση, εμείς χρησιμοποιούμε τα, ε, το εναπομείνον πλουτόνιο για ε, παραγωγή νέων καυσίμων το ανακυκλώνουμε ε, μέσα στο ίδιο το πυρηνικό εργοστάσιο, το αποθηκεύουμε και, όπως, ε, και προχωράμε σε ε, εκ νέου Λοιπόν, να σας δείξω λοιπόν αυτό το one-through αυτή την στρατηγική λοιπόν συνεχούς ροή, η οποία ακολουθεί πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές με αυτές τις ε, κάσκες τις οποίες έχει εγκρίνει και στη Βιέννη ο Διεθνής Οργανισμός ενέργεια, παρακολουθούνται όλα αυτά από το σημείο αναχώρησης μέχρι και το τέλος της μεταφοράς με τους παίκτες οι οποίοι ε, μπλέκονται σε αυτή τη μεταφορά που περνάνε από συνεχή επιμόρφωση, γυμνάσια και ασκήσεις. Μιλώντας λοιπόν για την κατάσταση και ποια είναι η στρατηγική ε, για την ανακύκλωση, να σας πω πως για την ιαλοποίηση χρησιμοποιούμε τις διάφορες τεχνολογίες που κυκλοφορούν στον πλανήτη μας. Μίλησα για τη Γαλλία, μίλησα και για το Ενωμένο Βασίλειο που χρησιμοποιεί την ίδια τεχνολογία στις εγκαταστάσεις στο Sellafield. Αυτή η στρατηγική εδώ και πολλά χρόνια χρησιμοποιείται ε, και στην Ιαπωνία, στο Ροκάσο Μούρα και μιλάμε εδώ για ανακύκλωση εξαντλημένου καυσίνου που θα χρησιμοποιηθεί στις εγκαταστάσεις στην Κίνα. Και αυτό που ακούμε πολύ συχνά, εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι πως η Ινδική στρατηγική ευθυγραμμίζεται με την Κινέζικη, δηλαδή ανακύκλωση ε, αναλωμένων καυσίμων. Μιλώντας για την τεχνολογία, θα ήθελα να μιλήσω πρώτα για την MOX τεχνολογία. Αυτή η τεχνολογία είναι το μεικτό οξύδιο που έχει ως σκοπό να διαχωρίσει το, πλουτόνιο που έρχεται από το στρατιωτικής χρήσης πλουτόνιο. Είπα και Ρωσία βασικές πηγές. Αυτή τη στιγμή στην Νότια Καρολίνα κατασκευάζεται μια τέτοια μονάδα και εκεί θα έχουμε παραγωγή MOX ε, από το, 20, από το 2016 για να χρησιμοποιηθεί σε πυρηνικούς πυρήνες ε, αντιδραστήρων στις Ηνωμένες Πολιτείες και χρησιμοποιούνται κάποια ε, πειραματικά συγκροτήματα απάρτια σε αυτές τις εγκαταστάσεις. Μιλώντας λοιπόν για τη διαδικασία η μιλάμε για μια διαδικασία στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης στη Γαλλία, στην Ιαπωνία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και που θα χρησιμοποιηθεί από την Κίνα και την Ινδία, αλλά πρέπει να σας πω πως η διαδικασία αυτή χρησιμοποιείται σε πολύ ραδιενεργά υγρά απόλυτα που προέρχονται από στρατιωτικά προγράμματα παλαιότερα. Είναι μια διαδικασία η οποία είναι στο εργαστήριο Savannah River για τη διαδικασία υλοποίησης με πολύ παλιά αποθεματοποίηση Programs. στα διάφορα προγράμματα εξάντλησης. Όταν μιλάμε όμως για ανακύκλωση, μιλάμε και για διαχείριση αποβλήτων. Όμως, παράλληλα, αναφερόμαστε και στη διαδικασία ανακύκλωσης, δηλαδή νέα χρήση παλαιότερων υλικών για παραγωγή ενέργεια. Στη διαφάνεια αυτή θα ήθελα να σα παρουσιάσω τι δύο ε, στρατηγικές στρατηγικέ και τι επιπτώσει που έχουν στον όγκο καυσίμων που πρέπει να αποθηκευτούν, όπω επίση και στην ε, ποσότητα ηλεκτρική ενέργεια που μπορεί να παραχθεί. Να σας πω τι γίνεται στην, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μιλήσω και για τα νέα σχέδια που έχουμε, τα οποία γνωρίζετε και να σας πω το τι θα γίνει το 2030 με τις δύο στρατηγηθείς που έχουμε, δηλαδή την άμεση διάθεση ή την ανακύκλωση. Για την άμεση διάθεση, direct disposal, να σας πω πως δεν έχουμε παραγωγή ενέργειας. Με το υλικό το οποίο απλώς διατίθεται σε με κάποιο είδους εναπόθεση ή αποθήκευση. Και εκεί χρειάζεται 250.000 κυβικά μέτρα αποθήκευσης αποβλήτων, συσκευασμένων αποβλήτων. Με τη δεύτερη διαδικασία, αν φανταστείτε πως πρέπει να ανακυκλώσουμε όλον αυτό τον όγκο, θα μπορούσαμε με αυτό να παράξουμε με το ε, ανακυκλωμένο υλικό και με αυτό το, τη διαδικασία MOX, 11.000 ε, τελοβατόρες, τεραβατόρες ε, ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή 15 χρόνια οικιακής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι σημαίνει αυτό. Και ο όγκος προς αποθήκευση ε, μειώνεται στους 50.000 κυβικούς ε, τόμους, δηλαδή καταλαβαίνετε πως γερούμε δια του 5 τον όγκο ε, ε, είναι κυβικά μέτρα, με συγχωρείτε, και αυτό σημαίνει ότι διαιρούμε δια του 5 τον όγκο που έχουμε παράξει κατά την άμεση διάθεση. Αυτή η διαδικασία λοιπόν εφαρμογής ε, χρειάζεται χρόνο. Ε, πήρα το παράδειγμα της Γαλλίας. Εμείς ξεκινήσαμε του παλαιού τύπου αποθήκευση την του 70. Η Εθνική, Εθνικός Φορέας ε, για την διάθεση της πυρηνικής ενέργειας δημιουργήθηκε το 1980. Λέγεται Άντρα και βλέπουμε πως όλη αυτή η προετοιμασία, ε, μελλοντική αποθήκευση ε, ε, πεπιεσμένου ή ελοποιημένου αποβλήτου προβλέπεται για το 2020-2025. Μιλάμε λοιπόν για 55 χρόνια από την αρχή, από την έναρξη αυτής της διαδικασίας. Είναι λοιπόν μια μακροπνοή διαδικασία και μακροπρόθεσμη διαδικασία η διαχείριση αποβλήτων με και γι' αυτό, ε, σύμφωνα με το δικό μας σκεπτικό, πρέπει πάντα να βλέπουμε μακριά και να κάνουμε κάποιες αναγωγές. Πιστεύουμε λοιπόν πως μια οδηγία για τη διαχείριση ραδιενεργών αποβλήτων και τη χρήση αυτών θα έφερνε πολλά πλεονεκτήματα. Γιατί θα παροτρύνει τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν ένα ασφαλές και βιώσιμο σύστημα διαχείρισης αυτών, θα συνεισφέρει στην ενίσχυση της ε, δημόσιας αποδοχής της πυρηνικής ενέργειας, θα συμπληρώσει το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο για να δούμε τι κάνουμε ε, με το, ε, τα πυρηνικά απόβλητα από τον πυρηνικό πυρήνα και θα προωθήσει το ευρωπαϊκό μοντέλο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο. Άρα λοιπόν, να σας κάνω μία σύνοψη και να σας τονίσω το εξή. Τι, ποια είναι τα θετικά πλεονεκτήματα που φέρνει η ε, ανακύκλωση. Μία εξοικονόμηση 25% φυσικού ουρανίου Δηλαδή με την ανακύκλωση αυτή και τη μετατροπή σε πλουτόνιο. Ε, αυτό για μένα είναι πολύ σημαντικό γιατί όλοι οι φυσικοί πόροι πρέπει να εξοικονομούνται. Πρέπει να τους εξοικονομήσουμε για τις μελλοντικέ γενναίες, α, όλους τους πόρους, ακόμα και το ουράνιο. Ξέρετε πως τα φυσικά στοιχεία και η εξοικονόμηση αυτών γενικά αυξάνει ε, τις τιμές Άρα λοιπόν τα υλικά αυτά, τα οποία προέρχονται από εξαντλημένα καύσιμα, μειώνουν τις τιμές που χρησιμοποιούν οι εγκαταστάσεις για την παραγωγή ενέργειας, με αποτέλεσμα να βλέπουμε ένα κόστος ανάκτησης και ανακύκλωσης, το οποίο είναι σταθερό, είναι ένα πάγιο κόστος και δεν ε, συμβαδίζει με τις διακυμάνσεις της τιμές φυσικού, φυσικού ουρανίου στην παγκόσμια αγορά. Άρα λοιπόν για τους πελάτες μας προσφέρουμε μία ε, τιμή η οποία Μιλήσαμε για μεταστοιχείωση σήμερα το πρωί, μιλήσαμε ε, για τους ε, επιταχυντές αντιδραστήρων και για την ε, γρήγορη παραγωγή. Όλα αυτά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην παράμετρο κόστους. Δεν μιλάμε για ένα σχέδιο. Εμείς εδώ και δεκαετίες εφαρμόζουμε αυτά που σας παρουσιάζω. Έχουμε βιομηχανική παραγωγή σε βιομηχανικές μονάδες, έχουμε εμπορική διάθεση, μιλήσαμε για το κόστος σήμερα το πρωί είναι πολύ χαμηλό το κόστος ε, και χαμηλότερο το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Άρα λοιπόν εμπορικά είμαστε ανταγωνιστικοί και βέβαια αυτή η ε, ανακύκλωση δίνει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον 10.000 θέσεις εργασίας, ε, σταθερές θέσεις εργασίας, αν λάβουμε υπόψη και τις υπεργολαβίες. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε πως στην οικονομία τη γενικότερη προσφέρει πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Και για την τελευταία αυτή διαφάνεια να σας πω και να σας υπενθυμίσω πως όλοι γνωρίζουμε την ανάγκη που έχει για ενέργεια, ηλεκτρική ενέργεια ο πλανήτης μας και προφανώς η ανανεώσιμη ενέργεια αποτελεί τμήμα της λύσης, όμως για εμάς είναι σαφές ότι και η πυρηνική ενέργεια αποτελεί τμήμα της λύσης. Η πυρηνική ενέργεια είναι μια ανακυκλώσιμη ενέργεια. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Ευχαριστώ και έτσι ολοκληρώσαμε ε, την ε, παροχή πληροφοριών ε, σχετικά με το θέμα αλλά δεν έληξε και η εκδήλωση και έχετε χρόνο να κάνετε ορισμένες ερωτήσεις αλλά παρακαλώ να είσαστε συγκεκριμένοι και σύντομοι για να μπορέσουν να απαντήσουν κιόλας οι ομιλητές. Ο κύριος Γκίρικ. την τεχνολογία KBS. Σε αυτά τα δοχεία από χαλκό η θερμοκρασία θα είναι αρκετά ψηλή φαντάζομαι. Επομένω, επομένως, αν το μέρος είναι απομονωμένο, ε, η θερμοκρασία μπορεί να ανέβει. Μετά από μερικά, μερικές εκατοντάδες χρόνια μπορεί η θερμοκρασία να ανέβει τόσο πολύ που να λιώσουν τα πάντα. Ε, και κάποια στιγμή να διαλυθεί απλώς ο μπεντονίτης από την υψηλή θερμοκρασία. Επομένως, δηλαδή, δεν θα είναι ο χώρος αυτός ε, σε θέση να λειτουργήσει. Επίσης, η ακτινοβολία Γ θα δημιουργήσει πρόβλημα στη δομή ε, του χαλκού και η διάβρωση θα είναι μια διαδικασία η οποία θα επιταχυνθεί. Υπάρχει τρόπος να παρακολουθήσουμε τις θερμοκρασίες σε αυτά τα δοχεία. Υπάρχει επίσης κάποιο σύστημα εξαρισμού, ούτως ώστε να ψήξουμε ε, το περιεχόμενο αυτών των δοχείων. Η κυρία Χάλμς, ε, δεύτερη ερώτηση. Έχω μία ερώτηση. Θα ήθελα να μου πείτε πώς είναι δυνατόν να υπάρξουν ε, τόσες αμφιβολίες για τη μέθοδο KBS και σε τόσες άλλες χώρες ε, συγχρόνως ε, προτιμάται το σουηδικό πρότυπο. Τι σημαίνει αυτή η συζήτηση στη Σουηδία για όλες τις άλλες χώρες οι οποίες ε, έχουν ακολουθήσει το Σουδικό πρότυπο χωρίς ε, να έχουν τα αναγκαία εχέγγυα και επίσης θα ε, ήθελα ε, να αναφερθώ εις το γαλλικό πρότυπο. Δηλαδή η Γάλλοι, η Αρέβα είναι σίγουροι ότι η επόμενη φάση όπου θα υπάρχει γρήγορη επεξεργασία θα είναι πιο επικερδής και αποτελεσματική από ότι η πρώτη που απέτυχε παταγωδός και η κατάσταση στη Γαλλία δεν είναι τέτοια σήμερα ώστε να πούμε ότι, το ε, ότι η ανακύκλωση πήγε τόσο καλά αλλά η Γαλλία είναι η χώρα όπου υπάρχει υπάρχει γενικώ ο μεγαλύτερος όγκος ραδιοενεργών αποβλήτων ε, στον κόσμο και όσον αφορά τον ε, κύριο Πατάκα αναφερθήκατε στο κόστος για την Φιλανδία όπου υπολογίσατε 100 χρόνια αν κατάλαβα καλά και μετά από 100 χρόνια ε, δεν θα έχετε πλέον κόστος για την ε, ε, εναπόθεση. Άλλες ερωτήσεις δεν βλέπω. Οπότε δίνω τώρα τον λόγο πρώτα στον κύριο Πατάκα ή στον άλλον ομιλητή πρώτα. Πώς, πώς θέλετε να προχωρήσουμε. Θα απαντήσω στα φιλανδικά. Να σχολιάσω ε, τα προβλήματα με τα δοχεία από χαλκό και τη μέθοδο KB, 3 ε, Η κατάσταση δεν είναι τέτοια που να οδηγήσει σε αύξηση της θερμοκρασίας αυτή τη στιγμή τοποθετήσουμε τα δοχεία μέσα στο πέτρωμα. Ε, μάλιστα η θερμοκρασία σύν το χρόνο θα κατέβει. Αν σας δείξω μάλιστα και κάποιους πίνακες, θα καταλάβετε ότι πρέπει να περιμένουμε δεκάδες χιλιάδες χρόνια ούτως ώστε να ψυχθεί αρκετά το περιεχόμενο των δοχείων ε, και μετά από 40 ή 50 χρόνια μπορούμε να περάσουμε στην τελική εναπόθεση. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν εμείς τι κάνουμε. ανακατεύουμε καύσιμο πιο θερμό και καύσιμο πιο ψυχρό. Ούτω ώστε το περίβλημα αυτό το, δοχείο που θα έχει, θα έχει 12 ράβδους καυσίμου, ψυχρούς ε, και ψυχρές και θερμές. Επίσης η θερμοκρασία έξω από το δοχείο δεν πρέπει να είναι πάνω από 100 βαθμούς Κελσίου. Αυτό είναι το σημείο αφετηρίας. Το θέμα τώρα το, του κόστους. Σας έδειξε ένα πίνακα με το συνολικό κόστος, τη συνολική δαπάνη. Και σας έδειξα και το χρονοδιάγραμμα. Μετά από 100 χρόνια, όπως σας είπα, θα κλείσουμε το χώρο αναπόθεσης. Ε, με βάση τη φιλανδική νομοθεσία υπάρχει η αρχή ότι θα πρέπει να σφραγιστεί το, ο χώρος αναπόθεσης και μετά η, ε, την ευθύνη θα την έχει το φιλανδικό κράτος. Θα περάσει δηλαδή από την εταιρεία Πόσιβα στο φιλανδικό κράτος, το οποίο θα είναι υπεύθυνο για το χώρο εναπόθεσης. Αλλά δεν πιστεύω ότι το κόστος ε, θα είναι ψηλό για την τελική εναπόθεση για τη διαχείριση της τελικής εναπόθεσης. Όταν κλείσει ε, ο χώρος αυτός, αφού κλείσει δεν χρειάζεται μετά ειδική επιτήρηση. Αυτό είναι σημαντικό για να ληφθεί υπόψη για το κόστος. Um, uh, Ο κύριος Πατράκα είπε σωστά ότι η θερμοκρασία δεν πρόκειται να αυξηθεί σε τέτοια επίπεδα που να δημιουργεί πρόβλημα και να λιώσουν ε, τα δοχεία αυτά χαλκού. Υπάρχουν τέτοια μοντέλα που θεωρούμε ότι μετά από λίγα χρόνια η εξωτερική θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 100 βαθμούς. Αλλιώς το νερό θα βράσει και θα, υπάρξει, θα όντως πρόβλημα. Αλλά γενικά η ιδέα με βάση τα μοντέλα είναι ότι η θερμοκρασία θα πέσει, θα είναι για 1.000 με 2.000 χρόνια ε, με, από 40 με 90 βαθμούς. Μετά θα επιταχυνθεί η διαδικασία διάβρωσης λόγω της θέρμανσης ε, του, χαλκού. Επίσης συζητάτε και το θέμα της ακτινοβολίας γάμα, της αδιανέργειας γάμα και πώς θα επηρεάσει αυτή το χαλκό. Ε, πριν από λίγες εβδομάδε ήμουν σε μια συνεδρίαση όπου ένας καθηγητής από τη Στοκχόλμη ζήτησε κάποιες εξηγήσει από την εταιρεία και Δεν νομίζω ότι ήταν ικανοποιητικέ αυτέ οι απαντήσει, αλλά τέλο πάντων ε, συζητείτε το θέμα. Δεν θα μετρηθεί η θερμοκρασία, δεν θα μετρηθεί η ακτινοβολία, ε, υπάρχουν συστήματα εξαιρισμού μόνο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, όχι όταν κλείσει ο χώρος εναπόθεσης. Αυτά για το χώρο εναπόθεσης. Ε, προς τη Ρεμπέκα Χάρμσα. πώς υπάρχουν τόσες αμφιβολίες για το σουηδικό μοντέλο. Είναι ενδιαφέρον αυτό το θέμα. Το σουηδικό μοντέλο και εγώ το θεωρώ ε, θετικό, αλλά και πολλοί άλλοι στη Σουηδία, εδώ και πολλά χρόνια. Ε, το περιβαλλοντικό ε, κίνημα, όταν άρχισε να δραστηριοποιείται πριν από έξι χρόνια, ε, θεωρούσε ότι θα πρέπει να ασχοληθούμε κυρίως με την εξέβρεση εναλλακτικών μεθόδων. Τα τελευταία όμως χρόνια νομίζω ότι ε, προκύπτουν σημαντικά θέματα, ιδίως σε σχέση με τη διάβρωση του χαλκού. Ίσως γιατί η Σουηδία είναι πολύ μικρή χώρα, το σύστημα είναι περιορισμένο ε, και λίγοι άνθρωποι δουλεύουν για αυτό το θέμα. Δεν υπάρχουν ανεξάρτητες ε, επιθεωρήσεις. Όλα τα λεφτά ε, για την έρευνα ε, πηγαίνουν σε αυτή την εταιρεία. Δεν, υπάρχει, δεν υπάρχει ανεξάρτητη έρευνα για αυτά τα θέματα στη Σουηδία. Ίσως λοιπόν υπάρχει μια προκατάληψη, ας πούμε, ένα είδος ιερατείο έχει δημιουργηθεί εκεί πέρα για αυτά τα θέματα. Και δεν έχουμε ανεξάρτητες δηλαδή έρευνες. Πάντως η βιομηχανία έχει όλη την ευθύνη ε, αν συμβαίνει αυτό, λοιπόν, θα πρέπει να έχουμε πολύ ισχυρέ ρυθμιστικέ αρχέ. Οι ρυθμιστικέ αρχέ θα πρέπει να μπορούν να ελέγχουν το τι κάνει η εταιρεία. Και ε, στη δεκαετία του 80 και 90 οι ρυθμιστικέ αρχές εξέταζαν μόνο τι έκανε η εταιρεία KBS και εξέταζαν τα αποτελέσματα για να δουν αν είναι απλώ σωστά. Δεν έψαχναν να δουν σε ποιους τομείς δεν κάνει έρευνα η KBS. Επίσης το θέμα της διάβρωσης του χαλκού έχει συζητηθεί. Ξεκίνησε στα τέλη της του 80 για πρώτη φορά, αλλά το ξεχάσαμε, το παραπέμψαμε στις καλένδες τότε και τώρα ανεφάνει τα τελευταία χρόνια. Τώρα το κόστος μετά την, το κλείσιμο του χώρου εναπόθεσης. Υπάρχει ένα κόστος το οποίο δεν λαμβάνουμε συχνά υπόψη. Στη Σουηδία το κράτος θα αναλάβει την ευθύνη για το χώρο εναπόθεσης μετά την πάση της λειτουργίας του, όπω γίνεται και σε πολλές χώρες. Όταν έχει τέτοιες, ε, τέτοιους χώρους ε, ε, εναπόθεσης αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου, έχουμε πλουτόνιο εκεί. Επομένω υπάρχει κίνδυνο εξάπλωση των πυρηνικών. Υπάρχει, θα πρέπει να υπάρχει λοιπόν κάποιο είδο παρακολούθηση. Η διεθνή κοινότητα θα πρέπει να έχει κάποιε ασφαλιστικέ δικλείδες για να εποπτεύει, να παρακολουθεί το χώρο. Αυτό θα πρέπει να είναι ένα θέμα που απασχολεί την κοινωνία μας. Ιστοδυναικές. Για χιλιάδες χρόνια η διεθνή κοινότητα θα πρέπει να επιτηρεί αυτούς τους χώρους εναπόθεσης. Υπάρχει κάποιο κόστος για αυτή την παρακολούθηση, αλλά δεν μπορούμε να μετρήσουμε με ακρίβεια ποιο θα είναι αυτό το κόστος της επιτήρησης των χώρων αυτών εναπόθεσης. Να δώσω το λόγο λοιπόν και στον τελευταίο ομιλητή, τον κύριο Χούγκελμαν, για να απαντήσει. Δύο βασικές ερωτήσεις άκουσα. Πρώτα απ' όλα, για την ιστορία του Super Phoenix, νομίζω αυτό ήταν το πρώτο, και δεύτερον για τον όγκο αποβλήτων που χρειάζεται να διαχειριστεί η Γαλλία. Καταρχήν, για το project αυτά, δεν θα πρέπει να σας δώσω πολλές λεπτομέρειες, γιατί το Super Phoenix είναι μια ιστορία που έχει να κάνει με την Υπηρεσία Κοινωνικής Οφελίας Παροχής Ενέργειας, στην EDF, και δεν νομίζω ότι μπορώ να δώσω ε, πολλές ε, λεπτομέρειες. Πρέπει να σας πω πως ε, ο παροπλισμός αυτής της μονάδας δεν ήταν μόνο τεχνικής δεν είναι μόνο προϊόν τεχνικής απόφασης αλλά και πολιτικής. Θα σας υπενθυμίσω μόνο πως εκείνη τη στιγμή το Phoenix που ήταν ο προκάτοχος του Super Phoenix λειτουργούσε πολύ ορθά και για πολλά χρόνια και παροπλίστηκε έκλεισε δηλαδή πριν από μερικά χρόνια μόλις. Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε ότι στο Phoenix και Super Phoenix ε, είχαμε παραγωγή MOX ε, τεχνολογίας, δηλαδή για την τεχνολογία τέταρτης γενεάς ε, για τους ταχύς αντιδραστήρες και για το Phoenix πρέπει να σας πω ότι ανακυκλώναμε ε, εξαντλημένα καύσιμα, αναλωμένα καύσιμα με τεχνολογία η οποία είναι πλήρως ε, συμμορφούται απόλυτα με την τεχνολογία που χρησιμοποιούμε για τους αντιδραστήρες ε, free breeder, τους επιταχυμένους. Πρέπει να σας πω πως είχαμε πολλές πληροφορίες, αποκτήσαμε πολλές γνώσεις για τέτοιου είδους αντιδραστήρες στη Γαλλία μέσω αυτών των μονάδων, οπότε αυτός εν μέρει απαντάει την ερώτησή σας. Δεν μπορώ να απαντήσω τίποτα άλλο παρά μόνο πω ήταν και τεχνικά και πολιτικά τα θέματα που προέκυψαν και οδήγησαν στο κλείσιμο. Δεύτερον, ανακύκλωση και διαχείριση αποβλήτων. Πρέπει να λάβετε υπόψη για, την, για τον όγκο αποβλήτων που διαχειριζόμαστε στη Γαλλία. Καταρχήν, τον όγκο της ε, ηλεκτρική ενέργεια που παράγουμε με, πυρηνικέ με ε, αναμεγαβατόρα ε, ή αναπυρηνικό αντιδραστήρα παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αν μιλάμε λοιπόν ανατόνο τόνο καυσίμου, ανά ή ανά εγκατάσταση, να σας πω πως η ανακύκλωση μειώνει κατά μειώνει πέντε φορές ε, την τελική ποσότητα πυρηνικών καυσίμων που πρέπει να διαχειριστούμε. Βέβαια, σε σχέση με τι περισσότερε χώρε, ο δικό μα όγκο αποβλήτων είναι τεράστιο, γιατί έχουμε τεράστια παραγωγή. Αν λοιπόν πυρηνική μονάδα ε, πολλαπλασιάσουμε ε, τον όγκο αποβλήτων και μετά το διαιρέσουμε με την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται, θα δείτε πως τα απόβλητά μας ε, δεν είναι τόσο εντυπωσιακά. Άρα λοιπόν εξαρτάται η διαχείριση των αποβλήτων από την τεχνολογία που χρησιμοποιείται και αυτή πολλαπλασιάζεται ε, με τον ε, όγκο της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται. Αυτές λοιπόν τις δύο παραμέτρους θα πρέπει να λάβετε υπόψη και να μην μιλάμε για απόλυτες συγκρίσεις σε όγκο αποβλήτων. Η Γαλλία δεν είναι η μόνη χώρα στον πλανήτη που παράγει πυρηνική ηλεκτρική ενέργεια α, ούτε είναι η χώρα που έχει τη μεγαλύτερη αποθήκευση αυτών. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι η χώρα αυτή και είναι μια χώρα στην οποία δεν έχουν κάνει την παραμικρή προσπάθεια ποτέ. Εγώ έχω ε, απαντήσει δίνοντα την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτείων. Βέβαια, ξέρω ότι εσεί θέλατε να εστιάσετε την ερώτησή σα στην Ευρώπη. Και θα πρέπει να θυμόμαστε πω αυτό ο όγκος ε, αντίστοιχων εγκαταστάσεων στην οποία αποθηκεύεται για την EDF όλο το ιαλοποιημένο συσκευασμένο απόβλητο υλικό. Μπορεί να γίνει στις 28 Ιανουαρίου και μπορείτε να πάτε εκεί να επισκεφτείτε την εγκατάσταση και να δείτε ε, τι ακριβώς γίνεται στη μονάδα, πώς αποθηκεύεται όλο αυτό το υλοποιημένο υλικό σκάσης, έτσι ώστε να διαπιστώσετε πως μιλάμε για μικρή ποσότητα, πολύ μικρό όγκο, ακόμα και αν είναι πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που παράγουν άλλα κράτη. Ωραία, ευχαριστώ. Η κυρία Χάρνς έχει ακόμη μία ερώτηση ε, σκέφτηκα ότι και σχετικά με τη Γαλλία η κατάσταση θα έπρεπε να παρουσιαστεί πιο συστηματικά διότι για την εργασία της Επιτροπής επί του θέματος αυτού είναι πολύ ενδιαφέρουσα η χώρα αυτή διότι η χρήση της ατομικής ενεργείας παίζει το μεγαλύτερο ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συγχρόνως διαπιστώνουμε ότι τα απόβλητα το οικονομικά απόβλητα που υπάρχουν τώρα στην Γαλλία μπορώ, δεν θα σας αναφέρω το κατάλογό μου αλλά μπορώ να σας τον δώσω στη συνέχεια μας αποδεικνύουν ότι υπάρχουν διάφορες ποσότητες διαφορετικών κατηγοριών αποβλήτων αλλά θα αναφέρω μόνο έναν αριθμό ο οποίος με τρόμαξε όταν ασχολήθηκα με το θέμα αυτό στη Γαλλία σχέση με τις άλλες χώρες δηλαδή αυτό που εγώ θεωρώ σαν ατομικά απόβλητα στη Γαλλία αντιπροσωπεύουν ε, αποθηκεύματα σε πάνω από χίλια σημεία εναποθήκευσης και ε, ε, ε, υπό πολύ υψηλές προϋποθέσεις ασφαλείας που πρέπει να υφίστανται όπως τονίζει ο, ο, ο Επίτροπος Έτιγκερ είναι αμφισβητήσιμο ότι αυτό όντως γίνεται έτσι στη Γαλλία και στη Γαλλία θα ήθελα να ξέρω εάν χρησιμοποιούν αυτές ε, τις τεχνικές που παρουσιάσαν οι συνομιλητές μας σήμερα. Διότι πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή στη Γαλλία τουλάχιστον δεν καλύπτονται αυτές οι προϋποθέσεις. Θέλετε εσείς να ξεκινήσετε. Νομίζω πως τα στοιχεία αυτά προέρχονται από το Εθνικό Πρόγραμμα Διαχείρισης ε, Αποβλήτων της Γαλλίας, το οποίο είναι ένα έγγραφο πολύ πλήρες με όλο τα πυρονικά απόβλητα που βρίσκονται στην εθνική επικράτεια και εδώ συμπεριλαμβάνουμε και τα νοσοκομεία, τις οδοντιατρικές ε, κλινικές που χρησιμοποιούν ακτινολογικό εξοπλισμό κτλ. Μιλάμε λοιπόν για χίλιους για χίλια σημεία συλλογή αποβλήτων. Ε, δεν έχουμε χίλιου πυρηνικού σταθμού. δεν έχουμε χίλιε μονάδε παραγωγή ε, ηλεκτρικής ενέργειας από πυρηνικά. Καταλαβαίνετε πω δεν είναι ε, πουδενή ε, χίλιοι, ε, είναι απλώ χίλια σημεία συλλογής. Ευχαριστώ για τις επιπρόκειτες διευκρινήσεις. Δεν βλέπω τώρα να υπάρχουν άλλες ανάγκες σχολιάσεως. Θα ήθελα να ζητήσω από όλους να μας ευχαριστήσουν. Μας βοήθησαν με τα δύσκολα θέματα και αυτό αποδεικνύει ότι εάν παρουσιάσει κανείς έξυπνα τα θέματα μπορεί ε, να έχει καλύτερες κριτικές και πιστεύω ότι όσοι έμειναν μέχρι το τέλος ήθελαν να γνωρίζουν όλες τις πτυχές της διαδικασίας σας.